Uh, uh, Α αρχίσουμε και όσοι αργήσουν άργησαν. Εμείς θα αρχίσουμε. Να καλωσορίσω καταρχήν τον Επίτροπο Χιωακίν Αλμούνια, ο οποίος θα μας κάνει μια εισαγωγή για τις τωρινές εργασίες που γίνονται για την πρόταση γίνονται και διαβουλεύσεις ε, ε, ε, διυπηρεσιακές που βρίσκονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι για την πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Μου δίνει την ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις σας πριν να περάσουμε στα τελευταία στάδια των συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα συμμετείχαν κατά την μακρά αυτή διαδικασία και τις συζητήσεις Εξετίμησα ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που αναλάβατε για να καταρτήσετε δική σας έκθεση που ήταν πολύ χρήσιμη σε μας κατά τις εργασίες αυτές. Όπως ξέρετε, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, για την περίοδο 2014-2020 είναι κομμάτι μια ευρύτερη στρατηγικής, των εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων που άρχισε από την Κομισιόν με δική μου πρωτοβουλία πέρσι το Μάιο. Αυτή, αυτός ο εξυγχρονισμός του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων αποσκοπεί στο να ευθυγραμμίσει καλύτερα το πλαίσιό μας για τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων με τους στόχους της στρατηγικής ανάπτυξης της, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και παράλληλα ε, θέλει σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές, σε όλες τις οδηγίες να εισαγάγει το στοιχείο του περιβάλλοντος. Όλες οι δημόσιες αρχές διαχειρίζονται ε, δημόσια κονδύλια των φορολογουμένων Ιδιαίτερα όμως τώρα που περνάμε σε, σε περίοδο εξυγίανσης μεσούσης της κρίσης πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα πώς χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τα δημόσια κονδύλια και πώς εξυπηρετούν έναν κοινό στόχο που αποφασίσαμε να θέσουμε για την έξοδο από την κρίση κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Επανέλαβα πολλές φορές ότι αυτή η στρατηγική εξυγχρονισμού αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις δημόσιες αρχές γενικότερα για να πετυχαίνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά με καλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα των επενδύσεων και να διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα πηγαίνουν σε επενδύσεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν λάβει χώρα χωρίς τις κρατικές ενισχύσεις και την ε, δημόσια αυτή υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά τις ε, περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές, οι αρχές αυτές αφορούν περιφέρειες στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αφορούν τις μειονεκτικές περιφέρειες στην Ευρώπη. Θέλουμε να προσφέρουμε πραγματική προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανάπτυξη αυτών των περιφερειών με τις εξυγχρονισμένες guidelines. Θέλουμε επίσης ε, να προλάβουμε ε, τον ανταγωνισμό των επιδοτήσεων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών ε, τώρα που ο προϋπολογισμός είναι στενός. Οι προϋπολογισμοί όλοι. Θέλουμε να ξυγχρονίσουμε τον τρόπο ανάλυση των έργων των επενδυτικών που καλύπτονται από τι κατευθυντήριε γραμμέ. Θέλουμε να εστιάσουμε το έργο τη Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού όταν αναλύονται τα έργα για να δηλωθεί η συμβατή ενίσχυση σε περιπτώσεις όπου είναι μεγάλα τα ποσά της ενίσχυσης και θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εσωτερική αγορά και να κάνουμε ευρύτερες εξαιρέσεις και να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ε, χρησιμοποιήσουν προγράμματα για, την, ε, για τις περιφερειακές ενισχύσεις συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές, ούτε, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να είναι απλούστερα τα συστήματα χειρισμού της ενίσχυσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρέπει να δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ε, επταετή υλοποίηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα έχουμε και ένα κανονισμό γενικό για τις ε, ε, εξαιρέσεις unblock γιατί πολλά θέματα θα τα χειριστούμε μέσα από τις εξαιρέσεις ε, τις ε, ευρύτερε. Δηλαδή δεν θα υπόκεινται σε κοινοποίηση εκ των προτέρων ε, στην Κομισιόν, αλλά θα καλύπτονται από τη συμβατότητα του προγράμματος στα πλαίσια του οποίου χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στις Βρυξέλλες θα πάρουν ενίσχυση στις περιφέρειες. Πολύ σύντομα τώρα να δούμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισάγουμε τώρα στις κατευθυντήριες γραμμές. Είχαμε υπόψη μας ε, όταν αλλάξαμε και εξυγχρονίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ζει σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Και όταν συζητούσαμε τις προηγούμενες guidelines πριν από 7 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν ένας προς τρία. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους ζούσε τότε σε περιφέρειες που καλύπτονταν από τις κατευθυντήριες γραμμές, τις guidelines. Τώρα είναι ένας στους τέσσερις. Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τα δυο πρώτα χρόνια της κρίσης, παρόλα αυτά και οι περιφερειακές ε, διαφορές, ανισότητες σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό που ζει σε αυτές τις μειονεκτικές περιοχές ε, ο πληθυσμός μειώθηκε οπότε έχουμε μια καλύτερη εξυγίανση της εσωτερικής αγοράς και αυτό το λάβαμε υπόψη κατά την κατάρτιση των νέων guidelines. Παράλληλα όμως αντιλαμβανόμεθα απολύτως ότι ζούμε μέσα σε μια πολύ βαθιά και σοβαρή κρίση. Ε, ενώ ο πληθυσμός που καλυπτόταν ήταν ε, το 45% πριν του συνόλου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα με το παρόν σχέδιο των περιφερειακών guidelines ο πληθυσμός που καλύπτεται σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 θα είναι 47,2%. Για τις φτωχότερες περιφέρειες ε, θα παραμείνουν οι ενισχύσεις στην ίδια ένταση, ενώ για όλες τις άλλες υποστηριζόμενες περιοχές ε, προτείνουμε γενικευμένη ε, μείωση της έντασης της ενίσχυσης επειδή θα πρέπει να αποφύγουμε ανταγωνισμό επιδοτήσεων και να, έχουμε, να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες διαχείρισης των δημοσιονομικών στις περιφέρειες που θα υπόκεινται στις guidelines. Ένα σημείο που συζητήθηκε επί μακρόν και θα συζητηθεί σίγουρα και εδώ μαζί σας είναι η πιο περιοριστική προσέγγιση στις ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων ε, στις λεγόμενες περιφέρειες C. Στις α περιφέρειες, κάτω από το 75% του κατακεφαλήνα έπτυσης Ένωσης, θα συνεχίσουμε να ε, έχουμε, να αντιμετωπίζουμε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και μεγάλες εταιρείες με τον ίδιο τρόπο, με χαμηλότερες, χαμηλότερη ένταση της ενίσχυσης σε σχέση με αυτή που έχουμε για τις ΜΜΕ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Στις περιφέρειες C θα είμαστε αυστηρότεροι, διότι θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα ε, του, του κινήτρου, η προστιθέμενη αξία της δημόσιας ενίσχυσης ε, ε, επενδύσεων από μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλότερη από την προστιθέμενη αξία που έχουμε αναλύσει και έχουμε δει να πραγματοποιείται όταν η ενίσχυση αυτή δίδεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφενός οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι επενδύσεις αυτών μπορούν να δηλώνονται βέβαια ε, Συμπατές και να ε, υποστηρίζονται με δημόσια χρήματα εάν συνάδουν με τις τομεακές guidelines, ενέργεια, περιβάλλον, έρευνα, καινοτομία, ε, κεφάλαιο κινδύνου. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις που είναι οι πιο σημαντικές guidelines σε ό,τι αφορά το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μαζί με τις περιφερειακές guidelines. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν guidelines ε, θέλουμε να ε, κάνουμε κάποιες αλλαγές εξυγχρονιστικές και πριν από το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να εγκρίνουμε guidelines για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και το κεφάλαιο κινδύνου και μάλλον και για τη guidelines για το περιβάλλον και την ενέργεια. Αυτές θα εγκριθούν στο τέλος, στην αρχή του επομένου έτους και σίγουρα πριν από τη θητεία αυτού του Κοινοβουλίου. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρξουν επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις που δεν θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της ενέργειας περιβάλλοντος ή το κεφαλαίου κινδύνου ε, ή τη έρευνα και το μία ε, ενέργεια και αν είναι σε περιφέρεια C πάνω από το 75% του ενωσιακού ΑΕΠ σε αυτή την περίπτωση Έχουμε κάνει πιο ευέλικτη την αρχική μας θέση και τώρα στην τελευταία εκδοχή των guidelines θεωρούμε ότι μπορούμε να δηλώσουμε συμβατή την ενίσχυση για να στηρίξει τις επενδύσεις αυτές με την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα γίνει σε καινούριε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε ε, που θα λειτουργούν ε, γιατί εδώ είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα που θα έχει το κίνητρο που θα δοθεί. Πρόκειται για νέα εγκατάσταση, για νέα επένδυση όπου δεν υπήρχε πριν τίποτε ή στην περίπτωση ε, υφιστάμενης εγκατάστασης επενδύσεις για ένα νέο προϊόν για να γίνει μια νέα γραμμή παραγωγής, όχι μόνο για να βελτιωθεί η υφιστάμενη εγκατάσταση. Παράλληλα στις κατευθυντήριες γραμμές, στις guidelines, όπως και στις άλλες guidelines της νέας γενεάς που στηρίζονται στη στρατηγική εξυγχρονισμού, θα ζητήσουμε πιο έντονη αξιολόγηση, ιδιαίτερα του αποτελέσματος του κινήτρου. Σε αυτές τις guidelines θα εισαγάγουμε ε, ρήτρες κατά της αλλαγής της έδρας, της μετεγκατάστασης, πιο αυστηρές από ότι τις παρούσες, θα κρατήσουμε τις παρούσες, και θα προσθέσουμε κι άλλες για να υπάρχει αντικίνητρο για κατάσταση, γιατί είχαμε την εμπειρία στο παρελθόν καμιά φορά οι επενδυτές ζητούσαν σε μια περιφέρεια ε, ενίσχυση και μετά έκλειναν το εργοστάσιο σε μια άλλη περιφέρεια ενώ είχαν τις ίδιες οι παρόμοιες δραστηριότητες έχοντας λάβει πολλές φορές ε, κρατική ενίσχυση. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας βέβαια τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών και των αραιοκατοικημένων περιοχών στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε στο βαθμό του δυνατού τον, ε, τις περιφερειακές ενισχύσεις και τις σχετικές guidelines με τις πολιτικές συνοχής και τις περιφερειακές πολιτικές. Επαναλαμβάνω εδώ και το έχω ξαναπεί πολλές φορές κατά τη διαδικασία αυτή ότι ο σκοπός των guidelines για τις περιφερειακές ενισχύσεις δεν μπορεί να είναι ευθυγραμμισμένος 100% με τις αρχές των διαρθρωτικών πολιτικών της Ένωσης. Ο σκοπός αυτής της υποστήριξης δεν ταυτίζεται ακριβώς με τους στόχους των περιφερειακών πολιτικών ή των πολιτικών συνοχής. Εκεί που χρειάζεται ευθυγράμμιση υπάρχει. Και εκεί όπου υπάρχει ανάγκη ε, απόκλησης από τις αρχές και αποδεικνύεται αυτό, ε, η παρέκκληση, η απόκληση δεν συνιστά πρόβλημα για μας. Είναι εύλογη, είναι αιτιολογημένη πολλές ως ένα βαθμό. Κυρία Πρόεδρε, αυτά ήταν τα βασικά που είχα να σας πω. Πριν μπούμε στη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα θέλαμε τώρα δεν ξέρω ποιος ε, θα ξεκινήσει. Θα ακολουθήσω τους κανόνες μας. Καταρχήν ο εισηγητής και μετά οι συντονιστές. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την προσέλευσή σας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ε, ε, Πρόεδρο. Ε, ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε στη συζήτηση αυτή και χαίρομαι γιατί στην εισαγωγή του είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια σχόλια από την πλευρά μου. Εγώ πρέπει να λάβω υπόψη μου τα πραγματικά στοιχεία. Τρία θέματα θα θίξω. Οι κρατικές ενισχύσεις ε, και η πολιτική συνοχής ε, παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. Υπάρχει δηλαδή μια, ένα πεδίο εντάσεων μεταξύ τους και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δεδομένα, τα σωστά δεδομένα για την ε, πολιτική συνοχής και τις περιφέρειες. Η ταξινόμηση των περιφερειών ε, στηρίζεται σε δεδομένα από το 2007 μέχρι το 2009 και εμείς Ε, έχουμε κάποια στοιχεία από το 2008 μέχρι το 2010 για τις περιφέρειες και έχουμε και τα στοιχεία για την ανεργία. Όλα αυτά δείχνουν μεγάλες διαφορές. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι δεν χρειάζεται να, ε, να, συνταυτίζονται τα δεδομένα μας. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ε, γιατί Χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση αλλά και μια απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιούχους. Φοβάμαι επίσης για το πώς ε, αντιμετωπίζομαι τα υποεθνικά όργανα στα κράτη-μέλη που αυτοί είναι που πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες ε, για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Πρόκειται για περιφερειακές διοικήσεις, ε, τοπικές ε, αυτοδιοικήσεις. Διοικήσεις που δεν, είναι, έχουν την απαραίτητη πείρα για να τα εφαρμόζουν όλα αυτά ε, και δεν θα μπορούν να εφαρμόζουν την πολιτική με τις απαραίτητες εξοικονομήσεις. Χρειάζεται λοιπόν ε, η υποστήριξη από την πολιτική συνοχή ε, για την οποία υπάρχει και ανάγκη κοινοποίηση. Νομίζω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούμε ότι οι διοικητικέ δαπάνες και η περιπλοκότητα όλων αυτών των διαδικασιών πρέπει να μειωθούν και όχι να αυξηθούν. Ε, αυτό είναι σημαντικό για να μην είναι οι πολιτικές μας αυτοανερούμενες και δεν εξυπηρετούν το στόχο. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια ε, και πολλοί διστάζουν να υποβάλουν αιτήσει. Και τώρα τα νέα σχέδια περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Επίσης, ε, η Κομισιόν δεν έλαβε τη σωστή απόφαση σχετικά με τον αποκλεισμό των μεγάλων επιχειρήσεων στην περιφέρεια, στις περιφέρειες ΣΕ. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα ε, σε μια εποχή όπου χρειαζόμαστε κίνητρα για την οικονομία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ή ε, ε, μάλλον κάνει μελέτες που μόνο εν μέρη πιάνουν το πρόβλημα. Πώς μπορεί να ε, να είχαμε πιο χαλαρούς κανόνες τις εποχές των παχιών αγελάδων όπου υπήρχαν ε, χρήματα και τώρα να κάνουμε το αντίθετο. Δεν μπορούμε δηλαδή με σούσεις της κρίσης να ε, έχουμε την πολυτέλεια μιας τέτοιας πολιτικής. Βέβαια με τα λόγια σας μετριάσατε λίγο την κατεύθυνση, την πολιτική έτσι όπως είχε αρχικά ε, παρουσιαστεί και αυτό πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Επίτροπε, δεν θα αναφερθώ σε ολόκληρη την έκθεση, αλλά θα ήθελα τέλος να πω ότι δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά το Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα συναπόφασης στην πολιτική συνοχή και ε, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ε, ενεργά την ε, νομοθεσία, ενώ από την άλλη πλευρά να ζητάμε μόνο κάποια σχέδια να τα αποσύρει η Κομισιόν. Αυτό είναι δημοκρατικό έλλειμμα και ελπίζω ότι σε εύθετο χρόνο θα διορθωθεί το πρόβλημα. Να πω επίσης ότι αυτές οι πιο ήπιες παρατηρήσεις που μετριάζουν το πρόβλημα είναι ευπρόσδεκτες. Και αν ενσωματωθούν στο σχέδιο τότε αυτό θα εξυπηρετήσει την πολιτική μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βλάσακ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα σημεία που θίξατε, χωρίς να μακρηγορήσω. Έτσι ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν και άλλοι. Καταρχήν, οι σχέσεις μεταξύ πολιτικής συνοχής και περιφερειακών κατευθυντηρίων γραμμών και τα στατιστικά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη. Είναι απόλυτα λογικό για τις περιφερειακές κατευθυντηρίες γραμμές να λάβουμε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δύο μήνες πριν περίπου για το 2010 και οι χαρτογραφήσεις της, ε, της ε, προηγούμενης ε, περίοδου δεν συνέπιπταν με τα διαρθρωτικά ταμεία. Βεβαίως οι χαρτογραφήσεις ήταν, προσέγγισαν αλλά δεν ήταν παρόμοιες. Ως προς το Leipzig Halle, πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές μετά την απόφαση της υπόθεσης Leipzig Halle. Η απόφαση του Leipzig Halle αναφέρει ότι πολλές φορές οι υπεύθυνοι των υποδομών, οι υποδομές έχουν μια οικονομική διάσταση που θα πρέπει να αναλυθεί από άποψη κρατικών ενισχύσεων και θα πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση χτες ήμουν στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού όπου συζητήσαμε τις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ άλλων και υποστήριξε το Συμβούλιο δύο κανονισμούς, δηλαδή τον κανονισμό ισχύως και τον ε, διαδικαστικό κανονισμό. Η τελική απόφαση επαφίεται στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο υποστήριξε γενικότερα την προσέγγιση του κανονισμού ισχύω, έτσι ώστε ανατομέα να δούμε τις κρατικές ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει ε, προηγούμενη ε, ε, προειδοποίηση προς την Κομισιόν. Άρα η Κομισιόν μπορεί να, να συμπεριλάβει περισσότερους τομείς στο, στο, στο πλαίσιο εξαιρέσεων συλλήβδιν εξαιρέσεων. Άρα μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτούς τους νέους τομείς με βάση τον καινούριο κανονισμό για να δούμε πώς θα εισαχθούν στην, στο πλαίσιο εξαιρέσεων, συλλογικών εξαιρέσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, υποδομές ευρυζωνικής. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις συλλογικές εξαιρέσεις κρατικών ενισχύσεων για την χρηματοδότηση υποδομών να τις δούμε μαζί με τις ε, ε, διαρθρωτικές κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα σε τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας, ευρυζωνικής κλπ. Θα δώσουμε τελική μορφή στις συζητήσεις μας ως προς την τομεακή αυτή προσέγγιση στο τέλος ε, του έτους, ως προς τα αεροδρόμια τώρα. Γίνεται συζήτηση γιατί το Leipzig Halle είναι αεροδρόμιο. Προωθούμε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις αερογραμμές με βάση τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. Άρα φύγεται ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να μπορούν να ε, χρηματοδοτούν τις υποδομές και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να ελέγχουμε τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη νέα γενεά κατευθυντηρίων γραμμών με βάση τα πλαίσια εξυγχρονισμού και με βάση την απόφαση Leipzig-Halle τη στιγμή που οι υπεύθυνοι υποδομών λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Ως προς τον διοικητικό φόρτο, συμφωνώ μαζί σας, εάν δείτε την εργασία που γίνεται για να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, βλέπετε πολλά στοιχεία απλοποίησης. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές με όλους τους ε, συνομιλητές μου το εξής. Όταν η Επιτροπή αναλύει μεγάλα προγράμματα με μεγάλα ποσά κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά για να, υπάρχει, υπάρχουν ίσοι κανόνες ε, δίκαιης πρόσβασης, έτσι ώστε να μην υπάρχει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και να προστατεύσουμε τους πολίτες που είναι φορολογούμενοι έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι γίνεται σωστή χρήση των ε, χρημάτων που καταβάλουν οι φορολογούμενοι με βάση τους στόχους που έχουμε αποφασίσει από κοινού και προσπαθώντας να είμαστε αποδοτικοί. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις των κινήτρων ή την καταλληλότητα της ενίσχυσης. Εάν υπάρχουν και άλλα μέσα, για να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο δημόσιο χρήμα, τότε θα τα υποστηρίξω. Αναφερθήκατε στις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα ίδια. Επίσης, ως προς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα ανταγωνιστικότητας και ανταγωνισμού και κρατικής ενίσχυσης, ξέρω ότι προτιμάτε την συναπόφαση και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, Συμφωνώ και θα είχα υποστηρίξει τη συναπόφαση. Μου είναι αρεστή, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω εγώ τις συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ. Μάνφρετ Βέμπερ. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτό που είπατε στο τέλος ότι εκτιμάτε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και θα, το υποστηρίξετε. Είναι σημαντικό αυτό. Και στην Ολομέλεια και εδώ ε, είχαμε μαζική προσέλευση που δείχνει ότι απασχολεί το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς. Ε, πρέπει όλοι να καταλάβουν πόσο δύσκολη είναι η ε, ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Αφενός θα πρέπει να ε, επιτρέπονται επενδύσεις, ε, να, δίδονται, ε, να δίδεται η δυνατότητα επενδύσεων στις περιφέρειες και από την άλλη θα πρέπει να απαγορεύσουμε την υπερβολική υποστήριξη στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, εκ μέρους του ΕΛΚ, κάποιες παρατηρήσεις. Τα, οι επενδύσεις για θέματα υποδομών. Αναφέρθηκε η αποφαση Λάιψη Χάλε και εμείς πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές διότι οι περιφέρειες θα έχουν νομική ασφάλεια. Θα υπάρχει δυνατότητα να προχωρούν στις επενδύσεις με νομική ασφάλεια και αυτό για τις θυγόμενες περιφέρειες είναι πολύ σημαντικό. Μην ε, τις σύρουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά. Γι' αυτό χαιρόμεθα που και στο Συμβούλιο ελήφθη η απόφαση αυτή. Τώρα, το μεγάλο κρίσιμο θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων και την ε, υποστήριξη, την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. Ε, φαντάζομαι ότι η μετεγκατάσταση είναι ένα πρόβλημα ε, γιατί αυτό πρέπει να απαγορεύεται αφού δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή αγορά ο περιορισμός ότι μπορούν να ενισχύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις όμως νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. Όταν μιλάμε για μειονεκτικές περιοχές είναι περιοχές, περιφέρειες ε, που χρειάζονται ιδιαίτερα τις βιομηχανικές συσπυρώσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν σας παρακολουθώ γιατί θα μπορεί να προωθηθεί ένα νέο προϊόν και μια, για ένα εντελώ καινούριο εργοστάσιο αλλά όταν σε μια μειονεκτική περιοχή ε, μια μεγάλη εγκατάσταση θέλει να εξυγχρονιστεί για να γίνει ανταγωνιστικότερη στο μέλλον, εκεί γιατί δηλαδή να μην μπορεί να βοηθηθούν με επενδύσεις. Σε αυτές τις περιοχές ε, χρειαζόμαστε αυτές τις βιομηχανικές εισπυρώσεις στα κλάστερ γιατί εξαρτώνται και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτές που αλλιώς δεν θα επιβιώσουν. Γι' αυτό ε, ε, λέω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείτε το θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ για τις κινήσεις που κάνατε μέχρι τώρα, μετακινηθήκατε στη θέση σας, αλλά ξαναδείτε αυτό το θέμα. Το ΕΛΚ επίσης θέλει 45% ανώτατο όριο με βάση τον πληθυσμό δηλαδή να ισχύσει το ποσοστό που ίσχυε δηλαδή μέχρι τώρα το 45% και τέλος να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, το θέμα της παγκόσμιας προοπτικής, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και λόγω της απελευθέρωσης των τελωνιακών διατάξεων, ε, έχουμε να κάνουμε με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Ποια θα είναι η εξέλιξη εδώ και πώς θα απαντήσουν οι νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την παγκόσμια τοποθέτησή μας. Και το δεύτερο για την περιφερειακή πολιτική, κατά το παρελθόν οι χάρτες μεταξύ περιφερειακών πολιτικών και ε, πολιτικών ενίσχυσης ε, δεν ταυτίζονταν. Ε, δεν ισχύει ότι θα πρέπει οι χάρτες αυτές να είναι παρόμοιοι γιατί υπάρχουν ορισμένες ε, περιφέρειες που πρέπει να ενισχυθούν και δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ε, ε, από την άλλη μπορεί να υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης χωρίς όμως να διατίθενται τα ποσά. Τέλος κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι που το είπα και στην Ολομέλεια και που με απασχολεί γιατί είμαι στην ε, περιφέρεια της Μεθορίου μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας και πρόκειται για τη διαφορά ε, που υπάρχει στο ποσοστό των ενισχύσεων. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σε παραμεθόριες περιοχές, ιδιαίτερα του πρώην σιδηρού παραπετάσματος, είναι εκείνοι που έπρεπε να κάνουν πολλά για την ε, ένωση της Ευρώπης στο Βερολίνο ή σε άλλες περιοχές. Δεν νιώθει κανείς τη διαφορά τόσο στις παραμεθόριες. Στο μέλλον λοιπόν θα μπορούσαν ε, να έχουν ε, ε, ορισμένες παραμεθόριες περιοχές ε, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, άλλες πολύ χαμηλό. Έχουμε ένα 25%. Εσείς προβλέψατε ότι το εθνικό επίπεδο, Βαρσοβία, Βερολίο, Βερολίνο, Βιέννη, Ρώμη θα μπορούν να αποφασίζουν και ε, ότι θα ε, μπορούν να ε, αντιμετωπίζονται ως προνομιακές περιοχές. Καλό είναι να, να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Οι πολίτες όμως αυτές τις περιοχές περιμένουν η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό επίπεδο να φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στις ενισχύσεις. Και οι υπεύθυνοι επιτόπου και οι πολίτες επιτόπου λένε ότι είναι ευρωπαϊκό καθήκον να διευκρινιστεί ότι δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από το 15% στις ενισχύσεις. Ίσως πρέπει να έχουμε ένα ειδικό πλαφόν για αυτές τις περιφέρειες που είναι ε, πολύ λίγες περιφέρειες, δεν είναι πολλές, αλλά ε, επομίστηκαν ένα μεγάλο κομμάτι της επανένωσης της Ευρώπης. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να εξεταστεί και αυτό και ενδεχομένως να συζητηθεί. Ε, ίσως υπάρχει απόφαση βέβαια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θα μπορούσε ίσως να επανεξεταστεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερ. Ήδη έχουμε συζητήσει πολλές φορές εμείς οι δύο αυτά τα θέματα, αλλά θα το κάνουμε και ενώπιον της Επιτροπής. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ήδη έχω πει τι σκέφτομαι, τι πρέπει να ενταχθεί στις κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε λάβει υπόψη και έχουμε αναλύσει και σταθμίσει όλα τα επιχειρήματα που έχουν εκτεθεί εδώ και ένα χρόνο διαπραγματεύσεων. Έχουν γίνει πολλές συνεδριάσεις ε, με συνομιλητές, κυβερνήσεις, κράτη-μέλη, περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και Περιφερειακών μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚΕ επίσης Είναι ένα κείμενο που με έχει απασχολήσει πολύ κατά τη διάρκεια της εννεαετούς θητείας μου πριν από την έγκρισή του. Νομίζω ότι η τρέχουσα εκδοχή του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών ασχολείται ιδιαίτερα με τις επενδύσεις για τις προς μεγάλες επιχειρήσεις. Το πλαίσιο είναι επαρκές κατά την άποψή μου και με βάση την ε, πείρα της Επιτροπής ως προς τις κρατικές ενισχύσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις και με βάση τις ε, μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ακαδημαϊκή έρευνα θα έπρεπε να αρκεστούμε στο αρχικό κείμενο, δηλαδή να ε, ορίσουμε την τομεακή προσέγγιση κρατικών ενισχύσεων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όμως πληθώρα απόψεων, κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι νέες επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις, greenfield ή νέα προϊόντα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παλαιότερες θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Δηλαδή προχωρήσαμε πέρα από αυτό που θα μπορούσαμε. Δεν μπορώ να κάνω άλλο βήμα και μη μου το ζητάτε, γιατί χρησιμοποιούμε δημόσιο χρήμα σε αυτούς τους δυσμενείς καιρούς. Εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επίτροπη, η οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τις κρατικές ενισχύσεις και έχουμε περάσει και τα όρια που μας έχουν τεθεί. Τώρα, ως προς τη σύμπτωση των χαρτογραφήσεων, εσείς μιλήσατε για τις όμορες περιοχές και το συνδέω, τα συνδέω αυτά τα δύο στη Βαβαρία. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν ορισμένες ζώνες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τρέχουσα χαρτογράφηση που θεωρούνται ε, περιοχές που λαμβάνουν ε, κρατικές ενισχύσεις γιατί είναι όμορες. Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο δεν θα είχαν συμπεριληφθεί και δεν θα μπορούσαν να είναι περιοχές ε, δικαιούχοι. Όμως στη χαρτογράφηση κινήτρων περιλαμβάνονται. Δηλαδή η χαρτογράφηση... Αυτογραφήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις δεν συμπίπτουν με εκείνες των διαρθρωτικών ταμείων που αφορούν τον συνάδελφό μου τον Γιωχάνες Χάν. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, η περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά τα μέσα μπορεί να είναι διαφορετικά, καθώς και η μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε προέβαλε μάλλον μία σύσταση. Εμείς βεβαίως έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Το ξέρω, ο κύριος Βέμπερ έχει ίσως λίγο διαφορετική γνώμη, αλλά τις κατευθυντήριες γραμμές τις ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ καλά κάνετε να προβάλλετε τις δικές σας προτιμήσεις ή δικαιώματα. Αλλά το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί του θέματος. Εγώ ε, έλαβα υπόψη τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν στις χαρτογραφήσεις ως προς τις όμορες ε, περιφέρειες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και δεν μπορούμε να δώσουμε διαφορετικές οδηγίες. Εγώ έχω μιλήσει μαζί σας και με άλλους Γερμανούς ε, συνομιλητές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και στο Bundestag ανέφερα πρόσφατα ότι αυτή η χαρτογράφηση θα πρέπει να ε, συμπληρωθεί από τη Γερμανία, από τις γερμανικές αρμόδιες αρχές. Και επειδή και εγώ ανήκω σε μια χώρα η οποία έχει σχεδόν ομοσπονδιακό χαρακτήρα, Ιωνί ομοσπονδιακό στη δική μου περίπτωση, ομοσπονδιακό στη δική σας, συμμερίζομαι την αρχή της επικουρικότητας που διέπει τις εργασίες μας και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει το δικό του κομμάτι. Η δική σας χαρτογράφηση αφορά αποκλειστικά τη Γερμανία. Γιατί αν ορίσουμε έναν γενικό κανόνα που να διέπει τους πάντες, ε, τότε εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα και όχι το Βερολίνο ως προς τις όμορες περιοχές, αλλά θα είχαμε 27 προβλήματα στη συνέχεια. Και θα ανοίγαμε πόρτες και παράθυρα εκεί όπου δεν υπάρχουν, με πληθώρα προβλημάτων. Από το 47 ε, και μετά υπάρχει και μία δημογραφική εξέλιξη στη Γερμανία και έχετε περιθώριο να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε παρά τη δημογραφική αυτή διόγκωση που υπάρχει. Ε, Λάμπερτ Βανίστερόι. Α, Κωνσταντσε, Κωνσταντσε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μιλάω μόνο συντονίστρια, αλλά εκπροσωπώ και την Μάρσα Κλέμπερ τη Σκιώδη συγκίτριά μας που δεν μπόρεσε δυστυχώς να έρθει σήμερα και με παρακάλεσε να προσθέσω κάποια πράγματα και εξ ονόματός της. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν ήδη οι συνάδελφοι, όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε πρώτο-πρώτο, ε, Επίτροπε Αλμούνια. Νομίζω ότι σωστό είναι να μιλάμε για αρμοδιότητες, ο καθένας δηλαδή πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει, αλλά στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να <clears throat> έχει ένα κοινό στόχο και προσανατολισμό. Την πολιτική συνοχής δεν την εφεύραμε για να προωθούμε εδώ και εκεί πράγματα. Εφεύραμε την ε, πολιτική συνοχή, ούτως ώστε οι περιφέρειες και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε μπροστά και να γίνουν ανταγωνιστικότερες. Και νομίζω ότι είναι θεμητό να έχουμε μία προσέγγιση που θα βλέπει τους χάρτες, την εδαφική κάλυψη δηλαδή το, της συνοχής ε, και των ενισχύσεων στο βαθμό του δυνατού. Και η προσέγγιση να λέμε ότι αυτό δεν τα είχαμε κάνει ποτέ, ε, αυτό τα ξέρω και από εκείνη την πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος γιατί μπορούσαμε να βλέπουμε τα σύνορα από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό σωστό είναι να προωθήσουμε περισσότερο και να ενισχύσουμε περισσότερο τις αδύναμες περιοχές, αλλά εξίσου σωστό είναι σε αναπτυγμένες περιφέρειες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην προωθούμε μόνο τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις μεγάλες. Και νομίζω ότι είναι ενδεδειγμένο αλλά αυτό είναι βέβαια δική σας αποκλειστική αρμοδιότητα, το αποτέλεσμα των δύσκολων διαπραγματεύσεων για το κανονισμό για τις περιφερειακές ενισχύσεις να δείτε ποιες ε, ε, εξαιρετικές ενισχύσεις ε, έχουμε συμφωνήσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν ε, άλλωστε δεν ε, ε, απέχει από το, τους τριμερείς διαλόγους, εκεί είναι και εκείνη. Κοινός μας στόχος και η πολιτική συνοχή έχει θέσει ως στόχο να προαγάγει την πολιτική Ευρώπη 2020. Κάνουμε δηλαδή ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε επιτυχίες στην επόμενη περίοδο. Καλό θα ήταν λοιπόν να επιδειχθεί μεγαλύτερη προθυμία, ούτως ώστε αυτή την ε, κατεύθυνση που την έχουμε ε, εγκρίνει και αναφέρει πολλές φορές και εδώ και στην Ολομέλεια. Ε, έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να σας ενθαρρύνουμε να δείτε μήπως μπορούν να υπάρξουν κάποιες σοβαρές τροποποιήσεις στην πρότασή σας. Επίσης κατάλαβα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια ότι είσαστε ανοιχτός για κάτι τέτοιο, να συμπεριληφθούν δηλαδή κάποιες βελτιώσεις στην ε, ρύθμιση για τις ενισχύσεις. Τώρα, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα γίνει αλλαγή στους κανόνες de minimis? Τώρα, στο γενικό κανονισμό, ε, είπαμε ότι ε, αν υπάρχει μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 10 χρόνια να είναι δυνατόν να απαιτούμε ανάκτηση χρημάτων που δόθηκαν ενισχύσεων. Ε, μια τέτοια ρύθμιση μπορείτε να προβλέψετε στις ρυθμίσεις περί ε, ενισχύσεων. Είπατε επίσης ότι θέλετε να προωθήσετε ιδιαίτερα τις νέες εγκαταστάσεις, ε, εντελώ καινούργιες. Τι γίνεται με την υποστήριξη και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που κάνουν αναδιάρθρωση ε, βιομηχανική και μπορεί να αλλάζουν κλάδο. Γιατί αυτό είναι μία επένδυση πάρα πολύ δαπανηρή και μας ενδιαφέρει αν θα πάρουν οι επιχειρήσεις εκεί μεγαλύτερη ενίσχυση γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο, δηλαδή ένα κίνητρο κατά της αναδιάρθρωσης, αν ισχύει η ενίσχυση μόνο εκ του μηδενός για νέες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, όπως είπα στην αρχή της εισήγησης μου, συμφωνώ ότι θα πρέπει να συγκλίνουμε στους ίδιους στόχους και συγκλίνουμε, δηλαδή ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις κρατικές ενισχύσεις. Μας διέπει μία και ενιαία στρατηγική, δηλαδή ο έλεγχος των ε, κρατικών ενισχύσεων και μας ενδιαφέρει να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα αυτό τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων με τους ε, γενικούς στόχους που έχουμε ορίσει στις γενικές μας ενωσιακές στρατηγικές. Γι' αυτό τα μείζωνα στα μείζωνα ζητήματα έχουμε παρόμοια προσέγγιση μέσα στα πλαίσια και μιας πολιτικής συνοχής που μας διέπει μέσω του ρυθμιστικού, ενιαίου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, των κανονισμών δηλαδή. Άρα, η μεταχείριση από τα ε, διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα από το ΕΤΠΑ, προτάθηκε από τον συνάδελφο Χάν και ήταν πιο ε, αυστηρή στρίκτο σένσου δηλαδή σε σχέση με τον κανονισμό που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στο τομέα της έρευνας και της καινοτομίας ή στον τομέα του ε, περιβάλλοντος και της ενέργειας. Τώρα το ΕΤΠΑ προβάλλει προγράμματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και με βάση τους στόχους μας υπέρ της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να ενταχθούν οι κρατικές ενισχύσεις και είμαστε συμβατοί με τις επενδύσεις προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Προχωρούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο εμείς, αλλά και το Ταμείο Συνοχής. μέσα στα πλαίσια του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχει σύμπτωση απόψεων σε σχέση με την αντιμετώπιση των μετεγκαταστάσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές κρατικών ενισχύσεων λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι όσοι μετεγκαθίστανται δεν λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις και είμαστε ακόμα πιο αυστηροί με τον νέο κανονισμό. Έτσι ώστε όποιος μετεγκαθίσταται να δούμε κατά πόσο λαμβάνει όχι οι κρατικές ενισχύσεις. Και αν ε, μία επιχείρηση έχει κλείσει μία μονάδα δύο χρόνια πριν από τη στιγμή που ζητά την ενίσχυση, τότε η περιφερειακή ενίσχυση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστεί ενδελεχώς. Και αν ο δικαιούχος ενίσχυσης μετεγκαθίσταται σε μία περιφέρεια υποενίσχυση και υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ μεταγκατάστασης και ε, περιφερικής βοήθειας, τότε η ενίσχυση δεν θα πρέπει να χορηγηθεί. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς τον ε, κανόνα de εκεί ορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ενίσχυσης. Δηλαδή κάτω από αυτό το κατόφλι, το de δεν χορηγείται ενίσχυση θα οριστεί το επίπεδο de μέχρι το τέλος του έτους. Εμείς όμως δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον κανόνα de minimis, με συγχωρείτε, και χθες στο Συμβούλιο υπήρξε σύμπτωση απόψεων επί του θέματος. Να μην αλλάξει δηλαδή αυτό το όριο de Και όσον αφορά τις ε, ξερέσεις ανακατηγορία διέπονται με βάση ένα συγκεκριμένο κανονισμό, ο οποίος ε, θα διευρύνει την ισχύ των ενισχύσεων που δεν χρειάζονται πρώτερη ε, κοινοποίηση. Είναι πολύ ε, λεπτό το ζήτημα, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στρεβλό στην εσωτερική αγορά, αλλάζοντας το όριο de minimis, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μάθαμε κάτι το πολύ σημαντικό με τον κανόνα de minimis, όταν αυξήθηκε αυτό το επίπεδο δύο χρόνια πριν. Είδαμε τι δυνατότητες δημιουργήθηκαν με αυτή την, από αυτή την άνοδο. Εδώ δεν μιλάμε για κατανομή χρήσης, αλλά για αύξηση του ορίου de minimis για αυτούς που χρειάζονται μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά. Εσείς αναφερθήκατε επίσης, όπως άκουσα, αναφερθήκατε στις επενδύσεις brownfield, δηλαδή βιομηχανικές, παλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Όταν μιλώ για greenfield, μιλώ για τον επενδυτή και για τη νέα μονάδα. Είτε πρόκειται για αγροτική περιοχή, είτε αστική περιοχή, βιομηχανική περιοχή. Δεν αναφέρομαι στο παρελθόν ή στη φύση της μονάδας ή του, της ζώνης αυτής, αν είναι αγροτική περιφέρεια ή όχι. Έχουμε 25 λεπτά και 5 ομιλητές, γι' αυτό θα αρχίσουμε το Herman Winkler. Έχουμε λίγο ε, καιρό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, καταρχήν ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας που τεκμηριώνουν την αφοσίωσή σας στο θέμα. Ε, Ευχαριστώ και για τις προσπάθειες που κάνετε να λάβετε υπόψη τις απόψεις μας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Εμείς ε, θεωρούμε το θέμα πολύ σημαντικό στην ε, Ανατολική Γερμανία γιατί ε, μας απασχολεί πολύ η διαφορά μεταξύ περιφερειών Α και Γ σε πολλές περιφέρειες δικές μας, Πόμεν, Μέκλενμπουργκ, στη Γερμανία ε, το θέμα είναι μεγάλο και θα ήταν σημαντικό οι χάρτες να ταυτίζονται όσο γίνεται περισσότερο. Όπως τα διαρθρωτικά ταμεία που είχαμε μεταβατικούς κανόνες θα μπορούσαμε να έχουμε και εδώ. Γιατί όχι. Γιατί να μην έχουμε σε μεταβατική περίοδο στα guidelines για τις περιφέρειες α και γ στο μέλλον, γιατί ε, επίσης ε, στις μεγάλες, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το καθοριστικό είναι ποιος ορίζει τι είναι το νέο προϊόν. Ένα παράδειγμα επίκαιρο που απασχολεί την Κομισιόν στη νάνο και στα νάνο και μικρο, μικροηλεκτρολογικά προϊόντα. Ε, Ε, όταν χρησιμοποιούνται ε, διαφορετικής διαμέτρου ε, πλάκες λιθίου για την παραγωγή ενός προϊόντος αυτό η αλλαγή συνιστά καινούριο προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό όμως για αυτό το τομέα της τεχνολογίας να ενισχυθεί η καινούρια παραγωγή. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν εγκαταστάσεις στην περιοχή Α με την πολιτική αυτή ε, απέναντι στις περιφέρειες Γ, αντίθετα θα παρατηρηθεί με την κατάσταση εκτός Ευρώπης. Οπότε σκεφτείτε το κι αυτό. Yes, uh, uh <clears throat> Κύριε εξετάζουμε όλοι μαζί το θέμα ε, της σχέσης μεταξύ των κατευθυντήρων γραμμών και της ε, πολιτικής συνοχής. Το δικό μου ερώτημα αφορά τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Είπατε ότι δεν είναι το ίδιο. Το θέμα όμως είναι αν αυτά τα δύο στοιχεία είναι συμπληρωματικά ή αν θα έπρεπε να είναι συμπληρωματικά. Γιατί έχουμε κάποια στοιχεία που επικαλύπτονται. Είναι κοινά, όχι συμπληρωματικά. Κοινά όμως, για παράδειγμα, εγώ είμαι για το ΕΤΠΑ. Το αναφέρατε προηγουμένως. Εκεί λοιπόν στο ΕΤΠΑ προσπαθούμε να αλλάξουμε το κείμενο με μια συγκεκριμένη πρόθεση. Για παράδειγμα, να δώσουμε τη δυνατότητα επενδύσεων πρώτον στις μεγάλες επιχειρήσεις και πράγματι συγκλίνουμε σε αυτά τα στοιχεία, όλο και περισσότερο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο της συνεργασίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι μόνο το πεδίο, αλλά και η μέθοδος λοιπόν. Υποθέτω ότι οι διαπραγματευτέ και οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή που θα συμμετάσχουν στον τριμερή διάλογο, αν προτείνουν κάτι, έχουν κατά νου τι κατευθυντήρε γραμμέ. Ή όχι. Γιατί δεν είναι οι ίδιοι. έρχονται να διαπραγματευτούν μαζί μα και παρουσιάζουν τι απόψει που θα ε, αντικατοπτριστούν στι κατευθυντήρε γραμμέ. Για να είμαστε ειλικρινεί, για μα δεν είναι σημαντικό ε, τι διαπραγματευόμαστε με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, αλλά με την Επιτροπή. Αυτό αυτός είναι ο μεγάλο θεσμό και το όργανο. Λοιπόν, με, μεγάλε επιχειρήσει. Δεύτερον, ενέργεια. Η πρόθεση είναι να επιτρέψουμε τη χρήση του ΕΤΠΑ σε επενδύσει στον τομέα τη ενέργεια, των μεταφορών. και της ε, κατανομής αποθήκευσης. Αυτή αυτό είναι το σχέδιο, αν θέλετε, να χρησιμοποιηθεί το έτυπα σε αυτόν τον κλάδο. Εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αν όμω με τι κατευθυντήριε γραμμέ δούμε ότι στον κανονισμό επιτρέπεται και στι κατευθυντήριε γραμμέ όχι, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Τρίτον, αερολιμένες. Εξετάζουμε λοιπόν ε, τη διαδικασία και το θέμα των ερωλημένων, ιδίω σε σχέση και με το περιβάλλον. Το τελικό στοιχείο αυτή τη στιγμή έχουμε επενδύσεις στους αερολιμένες εάν ε, ε, υπάρχει στοιχείο προστασίας του περιβάλλοντος. Ως εισηγητή. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερο, λοιπόν όταν διαπραγματεύομαι επί ενός στοιχείου αν αυτό θα αντικατοπτρίζεται ή θα συμπληρώνεται στις κατευθυντήριε γραμμές. Αλλιώς θα εκπλαγούμε αν μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων ε, δεν θα συνάδει, για να το πω διπλωματικά, ή ακόμα και θα αντίκειται στα όσα έχουμε διαπραγματευτεί. Και τελευταίο ερώτημα. Μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικό, ε, τι είναι αυτό Τη επίπτωση των κινήτρων, ο αντίκτυπο των κινήτρων. Γιατί αυτό καθορίζει για κατά πόσο είναι εφικτό να ξεκινήσει η επένδυση. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε λοιπόν πρακτικά ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των κατευθυντήριων γραμμών. Είναι ή δεν είναι συμπληρωματικά στοιχεία, συγκλίνουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ επιτροπών για την πολιτική. Πρόκειται για σύγκληση μεταξύ φορτικών πολιτικών. Ευχαριστώ. Υπήρξε και ε, η συμπαραγωγή και κάποια άλλα στοιχεία που αφορούσαν ε, τις υποδομές. Είναι σημαντικό στοιχείο. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Στο Στρασβούργο το συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε προέρχομαι από τη Μαδέρα που είναι άκρος απομακρυσμένη περιοχή και η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας φέρνει καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα τα συζήτησα μαζί σας διμερώς, δεν θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω τα ίδια. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση θα μιλήσω για τα καλά νέα. Ήδη γνωρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ως προς το καθεστώς που έχει αλλάξει για τις άκρος απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχουν 38 ε, μέτρα και για τα 26 δεν υπάρχει η πρόβλεψη της προγενέστερης προειδοποίησης το κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών δεν είναι απόλυτα σαφές για να δούμε ποια είναι, ποιο είναι το καθεστώς το οποίο δεν διέπεται από την προηγούμενη προειδοποίηση. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μία διασάφηση για να ξέρουμε ποια μέτρα δεν πρέπει να κοινοποιηθούν, καθώς επίσης και Γενικός Κανονισμός που διέπει αυτά τα καθεστώτα ανακατηγορία. Δεύτερον, μία παρατήρηση και όχι ερώτηση. Θα ήθελα να σταθώ στις κρατικές ενισχύσεις με μία φορολόγηση ε, που αφορά την περιοχή των Καναρίων, δηλαδή μια ειδική φορολόγηση για τις εισαγωγές εμπορευμάτων. Ισχύει μόνο, όχι μόνο για τα Κανάρια νησιά, αλλά και για τη Μαδέρα και για τις άκρος μακρισμένες περιοχές. Εσείς μιλήσατε για την ε, υπεράσπιση της εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα να προσέξετε αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα, διότι είναι ύψης της σημασίας ε, για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές δημιουργεί μια επιπλέον στρέβλωση της αγοράς στις εμπορικές συναλλαγές των δύο αυτών περιφερειών που δεν δικαιολογείται. Γιατί στον κατάλογο προϊόντων που ε, διέπονται από αυτό το καθεστώς εμπεριέχονται προϊόντα τα οποία ούτε καν παράγονται στα Κανάρια νησιά, γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο κατάλογος. Ευχαριστώ, ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που έθιξαν τα τρία αξιότιμα μέλη. Πρώτον, πώς ε, αντιμετωπίζουμε κάποιες ε, περιφέρειες σε μετάβαση. Έχουμε ορίσει ως ε, περιοχές γάμα, να το πω διαφορετικά μάλλον. Έχουμε θεσπίσει ως προκαθορισμένες περιοχές γάμα στις κρατητήρες γραμμές, χωρίς να περιμένουμε δηλαδή ε, τον ορισμό του εθνικού χάρτη, όλες τις περιοχές που με τα στοιχεία ε, του 2008-2010 έχουν ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που κατά την προηγούμενη περίοδο, 2007-2013, ήταν κάτω από αυτό το όριο. Ήταν περιοχές Α. Όλες οι περιοχές Α του υφιστάμενου κανονισμού που θα ξεπεράσουν το όριο τα επόμενα 7 χρόνια, το κατόφλι, θεωρούνται, προκαθορίζονται ως περιοχές γάμα. Σε άλλες ε, περιπτώσεις, οι άλλες περιφέρειες που δεν θα είναι περιοχές α και δεν θα προκαθοριστούν ως ε, περιοχές ε, περιφέρειας Γ και θέλουν να λάβουν ενισχύσεις στην επόμενη περίοδο, θα πρέπει να εξετάσουν την περίπτωσή τους όταν κάθε κράτος μέλος θα θέσει την εθνική του χαρτογράφηση. Και τα κράτη-μέλη που θα το κάνουν αυτό μέσα στους επόμενους μήνες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον πληθυσμό που διαμένει σε περιφέρειες Α και προκαθορισμένες περιφέρειες Γ ότι το όριο του πληθυσμού που ε, κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων που θεσπίζονται στα, στις κατευθυντήριες γραμμές και το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού θα πρέπει να κατανεμηθεί ε, στην επικράτεια αυτών των κρατών μελών με τις εθνικές τους διαδικασίες. Εκεί δεν παρεμβαίνουμε. Ελέγχουμε τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις περιφέρειες Α συν τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις προκαθορισμένες περιφέρειες Γ τις παλιές α που πλέον γίνονται γ. Η διαφορά πρέπει να συμπληρωθεί από τις εθνικές αποφάσεις μέχρι το όριο, την οροφή που έχει ε, θεσπιστεί για κάθε κράτος μέλος. Πώς ορίζουμε το νέο προϊόν. Αναφερθήκατε σε κάποια τεχνολογικά προϊόντα, ε, τα μικροτσίπια του που παράγεται στη χώρα σας. Τα συζητούσα με τη συνάδελφό μου Νέλη Κρούς και με τους συναδέλφους της και τη Γενική της Διεύθυνση και έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, ειδικά για αυτόν τον κλάδο. Έχουμε κοινή αντίληψη λοιπόν και ερμηνεία του όρου του νέου προϊόντος. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτός ο ακριβής ορισμός του νέου προϊόντος για να αιτιολογείται η συμβατότητα μιας ενίσχυσης επένδυσης σε μεγάλη επιχείρηση σε περιφέρεια Γ θα πρέπει να αναλύεται κατά περίπτωση από εμάς. Σε περίπτωση μεγάλων προγραμμάτων, όπως και να έχει, θα έχουμε σε βάθος ανάλυση της αιτιολόγησης που θα υποβληθεί και θα πρέπει εκεί να ορίσουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε και να βρούμε έναν γενικό κανόνα που θα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις σε κάποιε περιπτώσει θα πρέπει να τα εξετάζουμε πιο ενδελεχώς. Ε, Αλληλεπικαλύψεις. Όπως είπατε, είμαστε ε, ένα συμβούλιο επιτρόπων. Έχουμε εξαιρετικά καλές επαφές και συζητήσεις ε, με τον συνάδελφο Γιωχάνες Χάν και οι ομάδες μας, αν θέλετε, συμμετέχουν ε, και συνεργάζονται συνεχώς και οι γενικές μας διευθύνσεις Οι συνάδελφοι λοιπόν του Γιώχανες Χάν ούτε Γενική Διεύθυνση Περιφερειών δεν θα εκπλαγούν από την πορεία των συζητήσεων γιατί παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ ε, τις Εάν θέλετε ως εισηγητή για τον κανονισμό του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης πέραν των διασφαλίσεων μου ότι υπάρχει συντονισμό, να έχετε και για συγκεκριμένη συζήτηση για τις λεπτομέρειες των νέων κατευθυντήριων γραμμών βεβαίω, και, το, και η ομάδα μου αλλά και εγώ προσωπικά αν και δεν είμαι εμπειρογνώμων ε, και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μαζί και με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών είναι στη διάθεσή σας. Μπορώ να σας πω όμως ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα εκπλαγούμε. Πότε θέλετε να συναντηθείτε με την ομάδα μου στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί, το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα, όποτε θέλετε. Εγώ θα υποβάλω την, ε, την πρόταση για γενική ε, έγκριση των καθητήριων γραμμών στο Συμβούλιο των Επιτρόπων στα μέσα του Ιουνίου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν έχουμε χρόνο να ε, οργανώσουμε μια συζήτηση με τα χαράς. Για τον αντίκτυπο των κινήτρων μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτή τη συνάντηση για να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο ο αντίκτυπος κινήτρων. Έχουμε βέβαια τεχνικές ε, ανάλυσης ε, αυτού του αντικτύπου. Πρόκειται λοιπόν για την ανάλυση του αντίβαρου, αν θέλετε. Τι θα συμβεί αν δεν δοθεί η κρατική ενίσχυση με το ίδιο πρόγραμμα. Θα γίνει το πρόγραμμα, θα γίνει στο ίδιο μέρος, στην ίδια περιφέρεια, υπό τους ίδιους όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ε, δίδεται αντίκτυπος κινήτρου στο πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα δεν λάβει χώρα τελικά ή είναι εντελώ διαφορετικό ή γίνει σε διαφορετική περιοχή, περιφέρεια, ελλείψη κρατικής ενίσχυσης, και η κρατική ενίσχυση θα είναι το τελικό επιχείρημα που θα πείσει τον επενδυτή να πραγματοποιήσει ε, την επένδυση ή να την κατευθύνει προς αυτή τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Εκεί υπάρχει λοιπόν ζήτημα κινήτρου. Επομένω, μια τέτοια επένδυση Greenfield εξορισμού έχει τέτοιο ε, αντίκτυπο κινήτρου. Συγγνώμη. Όταν ο επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα σε αυτή την φάση. Όχι, δεν συνδέεται αυτό με αυτό το στοιχείο, συνδέεται με άλλη ρήτρα. Εκεί θα πρέπει να αποφασίσουμε σε επίπεδο επιτροπής τη συμβατότητα ε, μιας κρατικής ενίσχυσης και του προγράμματος ε, επένδυσης, αν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η καταβολή αυτό το πόρον δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν την ε, λήψη απόφασης. Αυτή είναι η ρήτρα standstill. Ο κύριος Τεξέιδα. Οι πλέον απομακρυσμένες περιοχές συζητήθηκαν αρκετές φορές και είπα εξ αρχής ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, περιφερειακής ενίσχυσης και ο ε, εξαίρεσης ανακατηγορία αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Στη μία περίπτωση χρειάζεται προγενέστερη ειδοποίηση ή κοινοποίηση, στην άλλη περίπτωση όχι, για να ισχύσουν ε, παραλλήλο. Θα ισχύσουν μάλλον παράλληλα. Ο κανονισμός εξαιρέσεων ανακατηγορία συζητείται, αλλά δεν θα εγκριθεί τον Ιούνιο, αλλά στο τέλος του έτους γιατί θα ε, εγκριθούν πριν από τις κρατικές ενισχύσεις, γιατί χρειάζονται χαρτογραφήσεις και χρειάζεται χρόνος για την κατάρτιση χαρτογραφήσεων. Θα πρέπει όμως να τεθούν σε ισχύ παράλληλα, διότι πρόκειται για τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Και στα Κανάρια νησιά μου έθεσαν το ίδιο ερώτημα και θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αναθεωρηθεί μέσα στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος που διέπει τα Κανάρια νησιά και τη Μαδέρα ή τις άλλες πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Χρειάζομαι όμως τη γνωμοδότηση του συναδέλφου μου Σεμέτα που ασχολείται με θέματα φορολόγησης από τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Εάν λοιπόν το θέμα αυτό των Καναρίων ε, συμμορφούται με το φορολογικό πλαίσιο, τότε έχει καλώς. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, τότε δεν μπορώ να χορηγήσω καμία ενίσχυση. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσω αυτή την ανάλυση ενδεχόμενης συμμόρφωσης ή μη με το φορολογικό καθεστώς. Η Μαρία ε, Ριγκόια Εντάχει, κύριε Επίτροπε, μετά από τις εξηγήσεις που μας δώσατε και επειδή μιλάμε για κατευθυντήριες γραμμές κρατικών ενισχύσεων, δεν μπορώ παρά να σας επιστήσω την προσοχή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις, περιφέρει... για τις περιφέρειες γάμα και για τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Θεωρείτε ότι αυτό δεν θα αποτελούσε πρόσκομα για τις όμορες περιοχές με τρίτες χώρες που δεν διέπονται σε κανέναν περιορισμό. Αυτή είναι η έκκλησή μου. Ξέρετε ότι αναφέρομαι στην Ανδαλουσία ιδιαίτερα. Η Μόνικα Χολμάιερ. Η κυρία Χολμάιερ. Μόνικα. Κάθομαι σε λάθος θέση, συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, εγώ είμαι από παραμεθόρια περιοχή με 250.000 κατοίκους και χάθηκαν το τελευταίο διάστημα 40.000 ε, θέσεις εργασίας που δεν δημιουργήθηκαν ξανά. Από το 2007 που μειώθηκε η διαφορά στις ενισχύσεις, εμείς είχαμε περίπου 25 με 30% διαφορά. Μετά είχαμε κατάρρευση της αγοράς εργασίας και από το 2007 η Κομισιόν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά αυτής της ενισχύσης και τώρα ε, δημιουργήθηκαν 27.000 θέσεις εργασίας πάλι. Μετά το 2007 ε, μπορέσαμε να διορθώσουμε κάπως τα πράγματα. Είπατε κυρία Αντιπρόεδρε ότι εσείς είστε ο αρμόδιος επίτροπος για, την, για τις κατευθυντήριες γραμμές. Όμως και η Κομισιόν συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνη για τη διαφορά στις ε, ε, ενισχύσεις. Ε, πάλι υπάρχει αυτή η διαφορά ε, του 25% στη δική μου περιφέρεια. Και δεν μιλάω μόνο για μένα, αλλά για όλες τις περιφέρειες που είναι εκτεθειμένες σε μεγάλη διαφορά. Ε, υπάρχουν και στην Αυστρία, όχι μόνο στη Γερμανία τέτοιες. Ε, είναι αυτοί που δεν είναι περιοχές Γ, αλλά είναι κοντά στις Α. Εμείς δώσαμε μάχη για να ανέβουμε λίγο περισσότερο. Ε, δεν είναι δίκαιο λοιπόν να λέτε ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσει η Γερμανία μέσα από την κατανομή των περιφερειών γιατί ε, αν μια παραμεθόρια περιφέρεια έχει γίνει ε, πιο ενισχυμένη και είναι σε ανταγωνισμό με μια βιομηχανικά αδύναμη περιοχή, τι θα κάνει η Γερμανία σε τελευταία ανάλυση. Θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό η Κομισιόν το προκάλεσε και αφού το προκάλεσε η Κομισιόν, εκείνη έχει και την ευθύνη να το λύσει, τέλος πάντων να συμβάλλει στην επίλυση. Δεν λέω να μην υπάρχει διαφορά όπως παλιότερα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχουμε διαφορά στις ενισχύσεις 25% και αναγνωρίζοντας ότι συνολικά γίνεται προσπάθεια να μειωθεί η διαφορά αυτή, όμως να ε, μας λέτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει γερμανικό πρόβλημα. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα να λάβετε λόγο και ο Άλμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε. Και εγώ είμαι από τη Βαβαρία, μια περιοχή που συνορεύει με την Τσεχία και μας χώριζαν 50 χρόνια τα σύρματα. Η ίδια κατάσταση όπως περιέγραψε η Μόνικα ε, υπάρχει και σε μας τα τελευταία 10 χρόνια 2.000 ε, από τους ε, περίπου 100.000 πήγαν στην Τσεχία. Και τώρα κατά την παραμεθό κατά μήκος της Μεθορίου ε, υπάρχουν πολλές ε, μεταναστευτικές κινήσεις. Ίσως ε, θα πρέπει στο, κατά, τη, κατά μήκος της, της Μεθορίου να μην είναι η διαφορά πάνω από 15%. Δεν λέω να, μην, να καταργηθεί, αλλά να μην υπερβαίνει το 15%. Αυτό θα ήταν υπέρ των θυγωμένων αν μας βοηθούσατε. Χαιρόμαστε που ε, τώρα δεν μας, χωρίζουν, ε, δεν χωρίζει η σύρμα, αλλά ε, θα πρέπει να μας χωρίζουν και μεγάλες διαφορές και εδώ μπορείτε να βοηθήσετε εσείς κύριε Επίτροπε. Για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι ενδογερμανικό το πρόβλημα και στο Στρασβούργο το συζητήσαμε και όσα Αυστριακή ε, από την κάτω Αυστρία θέλω και εγώ να προσυπογράψω τις ε, προτάσεις που, ε, που εκφράστηκαν. Διαφορά στις ενισχύσεις πάνω από 15% είναι απαράδεκτη. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα δώσω την ίδια απάντηση όπως και στους προηγούμενους ομιλητές. Όταν δείτε το παρόν κείμενο και τις κατευθυντήριες γραμμές, βλέπετε ότι μεταξύ μιας περιφέρειας ΣΕ που ορίζεται από τους κανονισμούς, που διέπεται από εθνικούς κανόνες, και με βάση μια όμορη περιοχή που είναι α, το ποσοστό που ισχύει είναι το 15%. Αυτή είναι η ποσοστή αναλογία που ορίζεται και εντάσσεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Χαίρομαι που συμπίπτουμε ως προς τις απόψεις μας και σε αυτό το σημείο. Και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι απάντησα στην κυρία Ιριγκόγια. Ε, ε, κυρία Κάρεμπαχ, Χολμάιερ, νομίζω ότι ε, απάντηση, αλλά κυρίως την κυρία Χολμάιερ θα ήθελα να πω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα ευθύνης. Ποιος ελέγχει τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Ποιος ορίζει την χατογράφηση του κάθε κράτους μέλους. Το κράτο μέλος. Το κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος και οι εμπλεκόμενες περιφέρειες. Ως προς την επικουρικότητα διαδραματίζει ε, με υψηλό ρόλο σε αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων και πολλοί από εσά το προανέφεραν αυτό. Εάν εγώ έλεγα ότι τα κράτη-μέλη δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη σύνταξη της χαρτογράφησης, τότε την ευθύνη θα την έφερε η Κομισιόν. Αυτό δεν θα σας άρεσε καθόλου. Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του και θα πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτό αφορά και τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι πρόκειται για μια δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων. Ευχαριστούμε κύριε Πέτροπε που μείνατε μαζί σας, ε, μαζί μας για μια μισή ώρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να θίξω δύο γενικά ζητήματα. Βεβαίως και γνωρίζουμε ότι τα χρήματα που επενδύονται μέσω αυτής της πολιτικής θα δαπανηθούν μέχρι το 2015 και ελπίζουμε η Επιτροπή να εξετάσει αυτό το ζήτημα και να μην ε, διαμορφώσει όρους γενικής αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τους κανόνες υπό τους οποίους ε, θα χειριστείτε τους ε, όρους κατανομής. Πρώτον. Δεύτερον, ελπίζω να κατανοείτε ότι προτιμούμε ε, περιφερειακούς, περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τις κλαδικές, γιατί η βασική αρχή της πολιτικής αυτής είναι ότι εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών, ενώ οι κλαδικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν μια ενιαία προσέγγιση για όλους είτε πρόκειται για τις υποδομές, ε, ενέργεια, για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα πράγματα είναι ίδια σε πολλές περιπτώσεις, ε, ανεξαρτήτως περιφέρειας. Ελπίζουμε λοιπόν να διατηρήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό ε, την περιφερειακή διάσταση στις κατευθυντήριες γραμμές γιατί έχετε και διαφορετικές διευθύνσεις για τα κλαδικά και τα περιφερειακά. Α, όχι, λέτε για να μην χάσουμε από τις περιφερειακές και τις γραμμές. Ε, κάτι τελευταίο και βεβαίως και σημειώνω ε, την παρατήρησή σας. Σας διαβεβαιώ ότι μερεμνούμε για την πλήρη συνοχή των αναλύσεών μας και των αποφάσεών μας χωρίς να ξεχνάμε ποτέ την περιφερειακή διάσταση ενός προγράμματος κρατικών ενισχύσεων. Ακόμα και αν Κάποια προγράμματα αναλύονται λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, προϋποθέσεις συμβατότητας ε, κλαδικού χαρακτήρα, το οποίο είναι λογικό βέβαια για την ενέργεια, για την ε, καινοτομία. Δεν μπορούμε εκεί να αξιολογήσουμε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα με διαφορετικά κριτήρια γιατί υπάρχει σε μία περιφέρεια ή στην όμορη περιφέρεια. Όμω, ε, βεβαίω και διασφαλίζουμε αυτή την ε, συνοχή και σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε, όπως είπα θέλουμε να υιοθετήσουμε στην Επιτροπή αυτές τι κατευθυντήριες γραμμέ τον Ιούνιο. Έτσι θα ξεκινήσει η διαδικασία ε, εθνικής χαρτογράφησης το δεύτερο εξάμεινο στα τέλη του έτους, αρχές 2014, θα έχουμε και τον Γενικό ε, Κανονισμό Εξαιρέσεων από την Επιτροπή και η πρόθεσή μου είναι να ε, εντάξουμε στο, στις κατευθυντήριες γραμμές ότι η θέση σε ισχύ των κατευθυντήριων γραμμών θα λάβει χώρα στα μέσα του 2014 για να υπάρξει και μια περίοδος ε, Ανάλυση εξηγήσεων, συζητήσεων για το περιεχόμενο των γραμμών για να αποφευθούν παρανοήσει ή για να τελειοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την, ε, το συντονισμό μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και των νέων κανονισμών των διαχρητικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Uh, to uh, ναι. Και εγώ συμπερασματικά να πω μόνο ότι αν κατάλαβα καλά θα περιμένετε την ψηφοφορία στα μέσα Ιουνίου της έκθεσής μου και θα την εντάξετε, θα εντάξετε κάποια στοιχεία στις κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως γι' αυτό. Η Επιτροπή πραγματικά εξετάζει συνεχώς ε, τις ε, εκθέσεις σας. Μην ανησυχείτε. Δεν ξέρω αν χειροκροτούμε για τους επιτρόπους, όχι. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στην παρουσία σας εδώ, κύριε. Ε? ε? Uh, Συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα για τις ψηφοφορίες. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα για δύο λεπτά να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση. Όπως γνωρίζετε, όσοι ήταν και χθε εδώ μαζί μας, δεν ήταν και τόσο, να το πούμε και αυτό. Γνωρίζετε ότι θέλουμε οι ψηφοφορίε για τους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς να λάβει χώρα στη συνάντηση του Ιουλίου για να οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να ξεκινήσουν και οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν να τελειώσει αυτό το ζήτημα μέχρι τον Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Η πολιτική αυτή θα τεθεί σε ισχύ στην 1η Ιανουαρίου. Αυτό εξαρτάται και από τις διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου με την Ιρλανδική Προεδρία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει συνδεθεί μέσω της εντολής μας και με τις διαπραγματεύσεις ε, των ε, δύο τροποποιήσεων του υφιστάμενου τίσου προπολογισμού. και στι πολιτικέ ομάδε και στι εθνικέ αντιπροσωπείε θα κάνετε τη συζήτηση αυτή για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον φετινό προπολογισμό και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική μα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι λοιπόν ε, να μην μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τι διαπραγματεύσει χωρί ε, να έχουμε τα τελικά στοιχεία ε, στο ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω της συναπόφασης. Θα ακούτε λογικά ότι δεν είναι σαφή αν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει για το ΠΔΠ μέχρι τον Ιούλιο. Είναι πιθανόν, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχιστούν και μετά το καλοκαίρι. Εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνο να μην υπάρξει ΠΔΠ. Και θα ήθελα να έχετε πλήρη επίγνωση των συνεπειών μιας τέτοια περίπτωση για την πολιτική μα για τι προσπάθειες των τελευταίων δύο ετών μπορώ να πω, γιατί υπήρξαν πολλές ε, ε, προκατακτικές ε, προσπάθειες για να προετοιμαστούμε για τις διαπραγματεύσεις και είχαμε και ένα πλήρες έτος διαπραγματεύσεων. Μπορεί να χάσουμε ε, τα αποτελέσματα αυτού του μόχθου μας αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΛΤΑΠΗ. Θα ήθελα να πω επίσης δεν επιμένω, δεν σας θέτω, δεν σας επιβάλλω κάτι. Απλώς να γνωρίζετε ότι υπάρχουν επιπτώσεις για την μη λήψη απόφασης για το πολιτεύθυνο νομικό πλαίσιο, για την πολιτική μα για το κατά πόσο θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου. Είναι προ συμφέρον λοιπόν να εξηγήσουμε και σε άλλου συναδέλφου που μπορεί να μην κατανοούν τι, ποια είναι η σημασία ε, του ετήσιου προπολογισμού για την πολιτική συνοχή, ότι σημαίνει θάνατος, ε, θάνατο για την πολιτική μα αν δεν έχουμε αυτή την πολιτική μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Αν λοιπόν μιλήσετε με κόσμο στις περιφέρειες και αυτοί ακόμα αυτό περιμένουν ακριβώς, να ξεκινήσει η πολιτική την 1η Ιανουαρίου. Σκεφτείτε το λοιπόν ότι η πολιτική αυτή χρειάζεται και ασφάλεια πόρων και χρηματοδότηση των συντηματών. Να ξεκινήσουμε τώρα την ε, ψηφοφορία. Παρακαλώ, εισάγετε τις κάρτες σας για να ελέγξουμε. Open the vote. Έναξη ψηφοφορία. What we have the list, the, the latest list. I hope. Okay, good. Uh, it works? Yeah. No, I think only if I can just sell. Τριάντα από τους 33 ενώ έχουν εισαχθεί 43 κάρτες. Κάποιοι λείπουν λοιπόν. Για νέους συναδέλφους να σας εξηγήσω ότι πρέπει να έχουμε μία ψηφοφορία εικονική για να ελέγξουμε. Απλώς εισάγετε τις κάρτες σας. Τέσσερις δεν έχουν ακόμα ελέγξει, τρεις. Ένταξη. Uh, on Έκθεση Ολτρικ Vlasak. Είναι η πρώτη έκθεση. Ας ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Κατά τμήματα, ζήτησε η Άλντε. Πρώτο τμήμα λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην οίκον 1. Όχι. Συμβιβαστική 2 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 8. Δεύτερο τμήμα. Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 και πάλι έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε τη συμβαστική 9, δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας, 21 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται με πολύ μικρή διαφορά, αλλά εγκρίνεται. Κάποιος ε, στάθηκε τυχερός. Τροπολογία 50. Ψηφορία κατά τμήματα και πάλι. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο, α, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Έκο, Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ. Ψηφίσαμε για την 100. Εγκρίθηκε, μην ανησυχείτε. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 κατά τμήματα και πάλι. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Καταπίπτει 107. Συμβουβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβουβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Α. Δεύτερο τμήμα της 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις ε, αναφορές, citations. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 5. Έναρξη. απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές απο... υιοθετείται. 7 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 8 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 9 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 11 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την 11, νομίζω ότι υιοθετείται. 11. Γιατί καταπίπτει? Η 11. Η 10 καταπίπτει. Νομίζω ότι έχω λάθος ε, λίστα ψηφοφορίας. Για την 11. Αυτό το αποτέλεσμα. Υιοθετήθηκε, εντάξει. Αιτιολογικές σκέψεις. <clears throat> Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Σωστά. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Α, τώρα δεν ξέρω. Καταπίπτει. 18 και 19 υπέρ. Από κοινού υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στις προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχουμε την αναφορική πρόταση 1 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 1. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 με 20. 2 υπέρ. Να ελέγξουμε και πάλι. Έναρξη. Και πάλι απορρίπτεται. Εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το β καταπίπτει. Ψηφίζουμε το 5. Employment 5 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και το 5. Suggestion 5 we check. The vote is closed. Ε, Ένα σοσιαλιστή παρακαλώ να βγάλει την κάρτα του, εντάξει, πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 19 υπέρ. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. We open for, suggestion 11. Έναρξη για την 11. The vote is closed. Πέρας. 22 κατά, 20 υπέρ. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε για την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. The vote is open. The vote is closed. Πέρας. And it's... Υιοθετείτε 33 υπέρ 6 κατά. Συγχαρητήρια. So now we go to budget 2014, Georgios Stavrakakis. Περνάμε τώρα στην επόμενη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 Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. So we go now to, no, to four, as I said. We go to four. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δύο υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αυτό. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη. Έρας. Υιοθετείται 41 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Σε χαρακτήρια Γιώργο. Να περάσουμε τώρα στη γνωμοδότηση του Ζαν Jacques ΣΕΠ για την στρατηγική τεχνολογία μεταφορών, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 6, υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 7. Έναρξη. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ, να ελέγξουμε τη 16, έναρξη. Πέρας. 17 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Περνάμε στην 17 υπέρ, Κατά. Αποχές. Νομίζω ε, ότι απαραίτητα θα σε ελέγξουμε. Πέρας. 20 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Δεν έπρεπε να είχα ελέγξει. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Συγγνώμη, Πέτρο, μπορεί να χάσει και πάλι όμως. 19 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. δεν είσαι τυχερό. 23 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του κυρίου Βλάσακ. Υπάρχει αρνητική ψήφο, Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 29 υπέρ να ελέγξουμε. Εντάξει. 14 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται, εντάξει. 29 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τα 29. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 με 15. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έναρξη. The vote is closed. Σαράντα μία ψήφι υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Ας περάσουμε στο σημείο 18 και πάλι έκθεση του κυρίου Βλάσακ για τον πολιτισμό και τις ε, δημιουργικές ε, επιχειρήσεις. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την 5 έναρξη. Πέρας. 21 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αναλέξουμε. πέρα. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε τη 15. Πέρας. Ισοψηφία, οπότε απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ να ελέγξουμε και τη 17 έναρξη πέρας απορρίπτεται 28 κατά συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, να ελέγξουμε το 32, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ, 19 κατά. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Έναρξη. Πέρας. 41 ψηφί υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην ογνωμοδότηση Μαρτίν Άντερσον. για την εφαρμογή της στρατηγικής για τους νέους. Υπάρχει προφορική τροπολογία για την 1. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Όσο έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Α εγκρίνεται. Τροπολογία 4 καταπίπτει. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται για τη 15 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 και πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Γάμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 να ελέγξουμε την 22. έναρξη. Πέρας. Και πάλι σου ψηφία. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Α. Και πάλι το ίδιο. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τερπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ να ελέγξουμε την 26. Άρχεται. Πέρας. Η 20 υπέρ, 22 κατά απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, έναρξη. That's it. Ε, Πέρας, 41 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Τελειώσαμε την ψηφοφορία. As Ας ε, συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μόικα, είσαι έτοιμη? Αγαπητοί συνάδελφοι, να αποχωρήσετε ήσυχα, ησύχω από την αίθουσα, παρακαλώ. Και αυτοί που θα παραμείνουν επίσης, σας ησυχάσουν. Uh, I would like to use maybe this time to inform also about the decisions made ε, θα ήθελα να σας ε, μιλήσω και για τις αποφάσεις των συντονιστών χτες για την ε, απόδοση των εκθέσεων. Το, οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές ανέλαβαν τον κανονισμό που προτείνει η Επιτροπή μετά την απόφαση του Συμβουλίου για τις διατάξεις σε σχέση με την χρηματοοικονομική ε, διαχείριση ε, χρημάτων από κράτη-μέλη που αντιμετωπίσουν ε, μεγάλες δυσκολίες. Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Σλοβενία και Κροατία στάλει επιστολή από την Προεδρία σε σχέση με την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή τη συνάντηση αυτή που έγινε, μάλλον πού θα γίνει με τα Εθνικά Κοινοβούλια φέτος στις 27 και 28 Νοεμβρίου. Αποφασίσαμε να συνεδριάσουμε λοιπόν τον Νοέμβριο 27 και 28 Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Ε, συζητήσαμε το θέμα και θα προτείνουμε, θα υποβάλουμε προτάσεις. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην τελική εκδοχή. Θα συζητήσουμε συζητήσουμε τις προκλήσεις εφαρμογής για την ε, επόμενη γενεά της πολιτικής συνοχής μετά από τη συνάντηση και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτής της συνάντησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης συμφωνήσαμε να μην αποστείλουμε επιστολή στους ε, διαπραγματευτές του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ζητώντας ε, ε, περισσότερες, περισσότερα κονδύλια για την περιφέρεια της Μαγιόρκα. Αυτή ήταν η απόφαση των, αυτές ήταν οι αποφάσεις των συντονιστών. Εγκρίνεται φαντάζομαι. Περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση της Μόικα κλέβα κέκους, εφαρμογή και αντίκτυπο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα πλαίσια της πολιτικής για τη συνοχή. Η κυρία Κέκους, καταρχήν έχω προετοιμάσει τα πάντα στα σλοβενικά γιατί νόμιζα ότι θα υπάρχει διερμηνία αλλά δεν προβλέπεται. Ζητώ συγγνώμη για τα όσχη και τόσο τέλεια ε, αγγλικά μου. Ελπίζω, ελπίζω την επόμενη φορά να, να υπάρχει διερμηνία. Χαίρομαι λοιπόν διότι σήμερα θα μιλήσουμε για την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την πολιτική συνοχής για να φτάσουμε σε ευφυή και συμπεριληπτική ε, ανάπτυξη, κάτι το οποίο έχει ε, αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις για την ε, συνολική μείωση της ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται στην στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτές οι πολιτικές προωθούν την ενεργητική, ενεργειακή με απόδοση και η πολιτική συνοχή είναι μία από αυτές προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται ε, βελτιώσεις ε, που είναι ε, ζωτικής σημασίας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτά ευεργετήματα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία απασχόλησης, ευκαιριών και ανάπτυξης ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής, ε, ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επίσης θα πρέπει να φτάσουμε στους στόχους ενεργειακής απόδοσης όπως είχαν οριστεί εκ των προτέρων ορίζοντας επιπτώσεις των μέτρων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε περαιτέρω αυτό το στόχο. Αυτό προσπαθώ να επιτύχω στην έκθεσή μου ε, η αυξημένη ενεργειακή απόδοση σημαίνει καλύτερες μεταφορές και πολιτικές στέγασης και κατασκευών. Επίσης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ο τομέας της στέγης αποτελεί κομβικό σημείο αυτής της έκθεσης. Προτείνω άμεσα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενεργειακής απόδοσης για την περίοδο 14-20. Έλαβα υπόψη τις ε, μελέτες για τις επιπτώσεις ε, του προγράμματος ή των προγραμμάτων με ε, ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδιαίτερα επειδή το ελεγκτικό συνέδριο λίγους μήνες πριν μας μίλησε για πολύ χαμηλή απόδοση. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ευθύς επενδύσεις με βάση τα ταμεία για την ενεργειακή απόδοση και είμαι πεπισμένη για κάτι τέτοιο. Υποστηρίζοντας την ενεργειακή απόδοση με επενδύσεις από τα διαφορετικά ταμεία κινούμαστε προς την ε, σωστή κατεύθυνση κατεύθυνση το, ο τριμερής διάλογος για τον ε, βασικό κανονισμό συνεχίζεται. Γι' αυτό δεν μπορώ να προδικάσω τα αποτελέσματα και τις λεπτομέρειες που θα συζητηθούν. Σήμερα λοιπόν προτρέχουμε κάπως και πιστεύω ότι μπορούμε να ενημερώσουμε αυτή την έκθεση με τροπολογίες που θα περιλάβουν ε, και τα δεδομένα της τελικής συμφωνίας από πλευράς ΕΤΠΑ και κοινού κανονισμού, βασικού κανονισμού. Θα υποβάλω και εγώ ε, μερικές τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την ε, ευαισθητοποίηση και διάδοση πληροφοριών, θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου το θέμα είναι ύψη της ε, σημασίας. Είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο ή ίσονο σημασίας, αλλά αφού μίλησα με τους εκπροσώπους περιφερειών και τοπικών αρχών, είμαι σίγουρη και ε, άκουσα ότι χρειάζονται καλύτερες πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες και καλύτερες για τις χρηστές πρακτικές, για τα ευεργετήματα από τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω νέων καινοτόμων επενδυτικών ε, μέσων. Τα επενδυτικά μέσα αποτελούν σημαντικό θέμα της έκθεσης. Θα θέλαμε περισσότερη εργασία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή μας έχει υποσχεθεί σε μας και τους εμπλεκόμενους φορείς χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα είναι έτοιμα πριν από την περίοδο προγραμματισμού, δηλαδή αυτή τη εβδομάδα ή το μήνα αυτό. Περνά ο χρόνος και δεν βλέπουμε πραγματικές προτάσεις. Εάν ε, λοιπόν θεωρούμε ότι οι διαχειριστικές αρχές θα εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια, τότε θα πρέπει να υπάρχει νομική σαφήνεια για να προετοιμαστούν. Δηλαδή λέμε τα ίδια που λέγαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Πιστεύουμε ότι τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καταστούν δυσχερή τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Και υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε νέους καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης. Τέλος, θα ήθελα να σας μιλήσω και για τον τομέα στέγασης γιατί η ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια αποτελεί το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εξοικονομήσεις ενέργειας στα κτίρια. Επίσης το Κοινοβούλιο σε διαπραγμάτευση με Επιτροπή και το Συμβούλιο μπόρεσε να ανταποκριθεί μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ ε, με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον ε, τομέα της στέγης. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να είναι ακόμα πιο δραστήρια και να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια του ε, καινοτόμου, ενός καινοτόμου οδικού χάρτη που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε επιχειρησιακά προγράμματα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που θα βοηθούσαν ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα. Στην έκθεση μιλώ για θέματα επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση και επικοδομητικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης. Νομίζω ότι είναι καλά τεκμηριωμένη η έκθεση και ε, πιστεύω ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία με τους σκιώδεις τον επόμενο μήνα. Ωραία. Αρχίζουμε με τους σκιώδεις. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω την κυρία Κλέβα Κέκους για την έκθεσή της και συμφωνώ με τις περισσότερες παρατηρήσεις της για τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και την ευαισθητοποίηση σχετικά με καινοτόμους πηγές και λύσεις ενεργειακές. Καλή είναι η νέα δημοσιονομική δήλωση που πρέπει να συνοδεύει τις παλιές ε, χρηματοδοτικές πηγές σε περίοδο κρίσης. Και διαβάζοντας την έκθεσή της είδα πολλά θετικά. Δεν θα τα αναπτύξω τώρα, απλώς θα αναφερθώ σε ορισμένα που βλέπω ίσως κάποιες αδυναμίες. Πρώτον, η λεπτή ισορροπία που βρέθηκε στις διαπραγματεύσεις για τους κανονισμούς για τη πολιτική συνοχή. Αυτή δεν πρέπει να διαταραχθεί από την έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ισορροπία. Επίσης, οι παρατηρήσεις μου δεν πρέπει να υπονομεύσουν την ισορροπία σχετικά με κάποιες τολμηρές δηλώσεις για την ενέργεια ή κάποιες ε, προϋποθέσεις που μπορεί να μην ισχύουν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Στη Ισκιώδης πρέπει να συζητήσουν λίγο τις παραγράφους 10 με 12 και υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης, των διαπραγματεύσεων και της ευελιξίας, αλλά αυτά μπορεί να λυθούν σε κάποιες χωριστές συναντήσεις η βασική μου ανησυχία είναι ότι μοιάζει σαν έκθεση από την Επιτροπή Ήτρα και όχι από την Επιτροπή Ρέτζη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή, ότι δεν συμφωνώ, αλλά της λείπει η ειδική, συγκεκριμένη περιφερειακή διάσταση που χαρακτηρίζει τη δική μας Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, πολλές παράγραφοι της έκθεσης ε, αναφέρουν και οι αναφορές για την ενεργειακή απόδοση είναι εκτός αρμοδιότητος αυτής της Επιτροπής. Εντάξει, μπορούμε να τις αφήσουμε, αλλά είναι πιθανό, αν μείνει το κείμενο όσο έχει, η Επιτροπή να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα ίσως, να πεθούν ζητήματα στην Ολομέλεια θα έλεγα κάθε πολιτική ομάδα να το εξετάσει με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Ήτρε ξανά το θέμα και μπορεί ίσω η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών να πάει λίγο πιο πίσω για να προλάβουμε. Αν αποφασίσουμε ότι δεν πειράζει και ότι δεν μας επηρεάζει αυτό, ε, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι έχει μια προτεραιότητα το θέμα. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις που μπορεί να θεωρηθούν παραπλανητικές σε σχέση με την οδηγία που εγκρίθηκε για την ενεργειακή απόδοση. Αλλά αυτό θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Τέλος, η έμφαση στην κλιματική αλλαγή αντί στο πώς μπορεί η ενεργειακή απόδοση να σώσει ε, τα χρήματα των φορολογουμένων μειώνοντας την καταλάλωση ενέργεια μου φαίνεται να είναι λάθος δεν εξυπηρετεί την προώθηση της ανεργιακής απόδοσης που είναι τόσο θετικό πράγμα. Ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι γνώμες μας για το κλίμα. Η έκθεση πρέπει να μείνει στο θέμα της και να μην θέσει ευρύτερους ε, στόχους σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και να μην αναφερθεί στα κλιματοϊκά. Πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο αντικείμενο της ίδιας της έκθεσης. Εκεί πρέπει να μείνει. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι αφού κάνουμε κάποιες αλλαγές και διορθώσεις θα είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση. Και θα ε, τη δεχτεί η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καρίμα δεν είναι εδώ. Ελίζαβε θα μιλήσεις εσύ. Λοιπόν, θα κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Γενική παρατήρηση. Η έκθεση πάει στη σωστή κατεύθυνση. Χαιρόμαστε για τις λεπτομέρειες που αναφέρει και που κρύβουν πολλή δουλειά και πολλές ε, ισορροπημένες και λεπτομερείς διατυπώσεις που δίνουν πολλά καλά επιχειρήματα. Αυτό μου αρέσει. Το αντικείμενο είναι δύσκολο και είναι δύσκολο να συνδυάσουμε τον κοινωνικό με τον οικολογικό παράγοντα και αυτό το κάνει στο κεφάλαιο 1 με τις γενικές παρατηρήσεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό Μάλλον εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτή είναι η περιφερειακή διάσταση. Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα και για τα χρηματοδοτικά μέσα. Συνδυασμός κοινωνικής και οικολογικής ε, διάστασης ε, και ε, αυτό είναι το βασικό που πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Πάντως η γενική κατεύθυνση είναι σωστή. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρομαι τα χρηματοδοτικά μέσα. Θα ήθελα επίσης να γίνει μια μικρή αναφορά στα υφιστάμενα μέσα που τα έχουμε ε, βάλει μπρος μετά την κρίση, το 4% που έχουμε στον τωρινό κανονισμό, γιατί είναι επιχείρημα πολύ στιβαρό, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο και στο μέλλον Κάποιοι θέλουν να είναι περισσότερο από το 4% στον παρόντα κανονισμό. Ε, αυτό δείχνει ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση διατηρώντας το. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που αναφέρεις στο σημείο 34 για το ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Εσύ ε, κάνεις μια παρατήρηση σχετικά με το τι έγινε, μπορούμε να μιλήσουμε και για τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι αυτό συνάδει με την έκθεση και την ε, διατύπωση που επιλέγεις. Αυτή είναι η μόνο παρατήρηση, γιατί τα επιχειρήματά σου είναι πολύ συνεκτικά και σαφή, περιεκτικά και σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ μεγάλη δουλειά που ανέλαβες και έκανες. Ευχαριστώ, Έντιτ. Άλλο συζητεί το λόγο. Ο με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Είμαι και στην Επιτροπή Ήτρε άλλωστε. Είμαι λίγο απογοητευμένη γιατί ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη σε εποχή οικονομικής κρίσης και ύφεσης δεν άδραξαν αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία για να κερδίσουν όλοι. Δημιουργούνται επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξης, εξοικονομήσεις. Και αυτό που λέει η Λίνα για περιφερειακή προσέγγιση είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να δημιουργήσουμε ευαισθητοποίηση η οποία χρειάζεται Και όπως λέει και η συγκήτρια, θα έχουμε τη μόχλευση που χρειάζεται για να έχουμε ε, συμπράξεις ε, ιδιωτικού και εξοικονομήσεις για την ενεργειακή, η ενεργειακή απόδοση είναι πολύ σημαντική αλλά και η οικονομική απόδοση και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο ίσως στην οικονομική απόδοση δηλαδή ιδιαίτερα μεσούσης της ύφεσης ή ε, μπορούμε να έχουμε εδώ οικονομικές αποδόσεις και για τα, σε ατομικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών και θα ήθελα να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να συντονιστούν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι πολίτες ε, τα θέλουν αυτά, είναι έτοιμοι και είναι θέμα πια ηγεσία ε, για να υπάρξουν οι δομές και να γίνουν όλα σε επίπεδο κοινοτή, ε, δήμων, περιφερειών κλπ. Και να επιτελεστεί καλή πρόοδος. Και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την καλή δουλειά και τη Λίνα. Πρέπει να συνεχίσουμε προς ταχώς. Γιατί είπαμε, θα υπάρξουν ωφέλη για όλους. Πολλά πράγματα βέβαια έχουν κόστος, τα ωφέλη μπορεί να είναι προσωρινά σε άλλες περιπτώσεις, αλλά εδώ νομίζω ότι θα συνεχιστούν να υπάρχουν ωφέλη για όλους και πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Λάμπερτ, εσύ ανέθεσες να ψηφίσει ο Σράνου για σένα. Για το τελευταίο θέλω να πω κάτι ε, που είπε ο κύριος Κέλλη για τον ανακυκλούμενο αυτό χαρακτήρα και αν ε, δαπανά κανείς χρήματα δεν είναι μόνο το ποσό των χρημάτων ε, σημαντικό και εσύ αναφέρεις τι έγινε τα τελευταία χρόνια σημαντικό είναι να έχουμε έσοδα και στην ενεργειακή απόδοση τα μέσα αυτά από την Τράπεζα Επενδύσεων οι νέες καινοτόμοι μέθοδοι χρηματοδότησης μπορεί να ε, ε, δώσουν πολύ μεγαλύτερη μόχλευση και τα παραδοτέα να είναι περισσότερα. Αν οι εταίροι ε, έρθουν με δικές τους επενδύσεις και υπάρχει συμφωνία ότι μετά από κάποια χρόνια όταν θα πληρώνεται λιγότερο, λιγότερο για τους λογαριασμούς ενέργειας τότε θα ξαναγυρίσουν τα κονδύλια στα ταμεία. Οπότε μπορούν πολλές ε, καταστάσεις να προκύψουν που δεν θα επηρεάζουν τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Και αυτό είναι καλό. Εμείς έχουμε πολλά περιφερειακά κονδύλια. για τους στόχους των ταμείων. Οι περιφέρειες που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους πρέπει να κάνουν τις δαπάνες αυτές. Αυτό το θετικό χαρτί πρέπει να το παίξουμε περισσότερο. Να μην θέσουμε περισσότερους στόχους, αλλά η Επιτροπή Ρέτζι είναι εξαιρετική επιτροπή για να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει και να δείξει ότι υπάρχει μόχλευση, γιατί εμείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συγκεντρώνουμε μαζί πολλούς παίκτες. Οπότε μπορούμε να θα σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Μπορεί να αυξηθούν οι τροπολογίες έτσι, είναι τώρα 27, μπορεί να γίνουν περισσότερες. Ο Γιάνν Όλμπριξ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για ένα τέτοιο κείμενο γιατί είτε θα παρουσιαστεί πριν από την τελική ψηφοφορία για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μόνο για να προωθήσει κάτι που θα γίνει αποδεκτό πρέπει να, κάνουμε, να προτείνουμε κάτι που έχουμε ήδη κάνει. Προτείνουμε δηλαδή ότι το έχουμε ήδη κάνει. Ίσως είναι καλύτερο να το κάνουμε μετά την αποδοχή, γιατί θα λέμε το, το χαιρετίζουμε αλλά είναι και η χρονική συγκυρία που είναι σημαντική λοιπόν. Ίσως είναι καλύτερο να το κάνουμε στη συνέχεια, μετά την ε, ψηφοφορία τον Ιούλιο, για να αποτελέσει τη βάση για το επόμενο βήμα μας. Δεύτερον, η παρατήρηση της Ελίζαμπεθ για το 4% είναι σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί δεν υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί ήταν ο επαναπραγματισμός που καθυστέρησε. Όχι επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ο αναπρογραμματισμός λοιπόν έγινε για το 4% σε ορισμένε περιπτώσει, αλλά πολύ συχνά είπαν ότι έχει γίνει ήδη γίνει, υποσχέθηκαν ε, τους πόρους, δεν τους χρησιμοποίησαν. Όχι δηλαδή να δείξουν ότι η αλλαγή είναι θετική και η ανταπόκριση αρνητική. Όχι, απλώς η αλλαγή καθυστέρησε να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Και τρίτον, στην περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να αναφερόμαστε και στη Σύνοδο των ε, Δημάρχων όχι μόνο ως ε, ένας πολύ ωραίος θεσμός, αλλά και σε ό,τι αφορά το έργο τους. Γιατί η Σύνοδος των Δημάρχων ε, είναι μια αρχή που προβλέπει ότι κάθε πόλη που θέλει να συμμετάσχει πρέπει να προετοιμάσει στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και το καθεξής. Αν δεν προετοιμάσουν το σχέδιο, δεν θα συμμετάσχουν. Αν προετοιμάσουν το σχέδιο, και αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια ταχεία διαδικασία, γιατί ξοδεύουν πολύ χρόνο και χρήμα για να προετοιμάσουν το σχέδιο και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει εμεί ω ε, Επιτροπή Ρέτζι να προετοιμάσουμε αυτή τη σύνδεση και να πούμε στα κράτη-μέλη ότι αν επενδύσουν στο σχέδιο θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση αν πούμε ότι στην εφαρμογή του ΕΤΠΑ, για παράδειγμα, στο Ταμείο συνοχή, οι πόλεις που έχουν προετοιμάσει το σχέδιο θα ακολουθήσουν αυτή την ταχεία διαδικασία, θα είναι κάτι χρήσιμο, ε, πρακτικό, που θα συνδέεται ήδη με την Επιτροπή Ρέτζι. Ευχαριστούμε, Γιώργη Μτσέλερ. Ähm, ναι. Να, δεν ε, θέλω να διαφωνήσω με τον συντονιστή, αλλά όταν μιλάει για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ε, ε, και ότι θα επανέλθουν, θα ανακτηθούν χρήματα. Αυτό αγαπητέ μου Λάμπερτ σπάνια συμβαίνει. Στο τομέα των κτηρίων είχαμε πάρει μέτρα ενεργειακή απόδοση για να περιορίσουμε το κόστο όμω, γιατί εν μεταξύ τιμέ ενέργεια είναι τόσο ψηλά που δεν γυρίζει πίσω ούτε σεντ. Ε, πάντως, ε, καλό είναι που η ενεργειακή απόδοση γίνεται από εμά κεντρικό ζήτημα. Οι κοινότητε όμω που πρέπει να πάρουν μέτρα ενεργικής λιτότητας και ενεργικής απόδοσης θέλουν να κάνουν εξοικονομήσεις για να επιτευχθούν και οι κλιματικοί στόχοι. Πολλές φορές όμως ε, είναι πολύ μεγάλο το βάρος που επομίζονται σε τοπικό επίπεδο και γι' αυτό πρέπει να παρέμβει η ευρωπαϊκή πολιτική ενισχύσεων. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και το στόχο τα κόστη που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στον τομέα της ενέργειας να περιοριστούν. Χωρίς την ψευδέστηση όμως ότι θα εξοικονομηθούν και κάποια, δηλαδή ότι θα γυρίσουν πίσω κάποια λεφτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως ε, οι επενδύσεις γίνονται για τον περιορισμό του κόστους και για να επιτευχθούν γενικότεροι στόχοι. Η πολιτική των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτό πρέπει να βοηθάει τις περιφέρειες και τους Δήμους όχι, δεν συμφωνώ, λέει ο κύριο Λάμπερτ. Γι' αυτό ζητώ το λόγο. Επειδή δεν συμφωνώ. Μπορεί να μην τα παίρνουμε πάντα πίσω τα λεφτά, αλλά η δυνατότητα υπάρχει. Πολλές, ε, σε πολλές επενδύσεις. Εάν δώσουμε μια επιδότηση, αυτή χάνεται. Εγώ θέλω στον τομέα ενεργειακής απόδοσης, όχι παντού, αλλά σε πολλές από αυτές τις επενδύσεις, μια δέσμευση να υπάρχει ότι εντάξει, οι τιμέ αυξάνονται, αυτό είναι άλλο. Ε, είναι η αγορά, είναι η πολιτική ενέργεια, αλλά μπορεί να υπάρξει μια δέσμευση. Τα χρήματα που δεν θα χρειαστεί να τα δαπανίσουν, γιατί θα έχει αυξηθεί η απόδοση, να γυρίσουν πίσω. Αυτή η προσέγγιση χρειάζεται και αν ανέβουν οι τιμές. Δεν μπορεί να δίνουμε λεφτά και τίποτε άλλο. Στο μυαλό μου πρέπει να υπάρχει και το στοιχείο του κέρδους, δηλαδή κάτι να βγάλουμε. Τώρα πρέπει να διαφωνήσω εγώ. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε, ας πούμε, στο μέλλον πώς ε, οι οδηγίες αναθέσεων θα ε, ε, καταρτίζονται. Διότι πολλές φορές λέμε ότι η χαμηλότερη προσφορά είναι η καλύτερη και όχι η οικονομικά και μακροπρόθεσμα πιο προσοδοφόρα. Παράδειγμα, στο Βερολίνο υπάρχει μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει ασανσέρ και υποδομές για κτίρια. Και εντωμεταξύ έκανε παγκοσμίω την καλύτερη προσφορά με ανάκτηση ενέργειας από την κίνηση των ασανσέρ κλπ. Αλλά όμως προσέκρουσαν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ε, σε άλλες εταιρείες που είναι πιο... και, είναι... και ε, ε, η δικιά μας είναι πιο ακριβή. Οπότε πολύ πιθανό είναι να μην προτιμηθούν τα δικά τους τα σανσέρια, οι ανελκυστήρες, αλλά να πάνε σε χαμηλότερες προσφορές που όμως θα αποδειχθούν πιο ακριβές όταν μπουν σε λειτουργία στο κτίριο αφού θα καταναλώνουν πιο πολύ ενέργεια. Ποιος θα αγοράσει τους ανελκυστήρες λιγότερες ευρωπαϊκές οικοδομές ή μεγάλοι επενδύσεις. Οι Κινέζοι αγοράζουν αυτούς τους ανελκυστήρες ε, γιατί φαίνεται ότι έχουν πιο μακροπρόθεσμη πολιτική. Καλό είναι λοιπόν να δούμε και εμείς τον τρόπο σκέψης μας εδώ. Ναι, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι στο ΑΕΛ πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις. Οι πολιτικές ομάδες πρέπει να κάνουν ουσιαστικές συζητήσεις. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορείτε να αναφερθείτε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και τι πρέπει να γίνει, αν πρέπει να ανασταλεί, να αναβληθεί η ψηφοφορία ή να καταλήξουμε σε μια άλλη διατύπωση. Ναι, αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Εξ αρχής, αυτή ήταν η πρόθεσή μου να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε υπάρχει στις διαπραγματεύσει και συμφωνηθεί. Δεν έχει νόημα να έχουμε έκθεση που δεν θα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα Χρειάζομαι όμως και βοήθεια από τη γραμματεία. Θα, αν ψηφιστεί το Σεπτέμβριο, αν υπάρχει δυνατότητα, τον Ιούλιο. Εκτός μικροφώνου μιλάει πρόεδρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα τον Ιούλιο εξαιτίας του Γενικού Κανονισμού. Τέλεια. Ναι, αυτή την πρόθεση είχα και με τις τροπολογίε, γιατί προ το παρόν έχουμε ένα γενικό κείμενο και μετά θα έχουμε τις τροπολογίε βάσει των διαπραγματεύσεων. Να προτείνω το εξή. Έχουμε ε, προθεσμία στι 11 Ιουλίου, Ιουνίου, διορθώνει πρόεδρο, για τις τροπολογίε, Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα για την εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων και Υπάρχουν και συζητήσεις με την Ήτρε για τα ΕΦΗ e e δίκτυα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και εκεί για να μην ε, φέρουν μετά μια άλλη τροπολογία στην Ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν την προθεσμία υποβολής καταθέσεων μέχρι τις 11 ε, Ιουνίου. Μπορούμε λοιπόν ε, να δούμε τι θα γίνει και με τις διαπραγματεύσεις και να δεις και εσύ αν μπορείς να καταλήξεις κάπου. Υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση. Ποτέ δεν είναι βαρετή. Χάρη στο ΕΛΚ, πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Ναι, μάλλον πρέπει να τα συζητήσουν ε, στο ιστορικό του ΕΛΚ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που πήρατε το λόγο. Θα προσπαθήσω, γιατί εξ αρχής ήξερα ότι έπρεπε να αφήσω ένα χώρο ε, για την υποβολή τροπολογιών. Σίγουρα οι προτάσεις σας θα είναι εξαιρετικές. Άκουσα πολύ καλές προτάσεις και είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με απασχόλησαν στην αρχή στο Κοινοβούλιο ήταν τα μη προτιμησιακά μέσα και όπου υπήρχε δυνατότητα προσπάθησα να το αξιοποιήσω. πιστεύω πολύ στον ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων ε, ως ε, τρόπο προώθησης ε, της πολιτικής μας. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας. Με τις τροπολογίες δεν περιμένω κάτι πολύ σύντομα. Σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τον Ιούλιο. Ωραία. 11 Ιουνίου λοιπόν στις 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ε, υποβολή τροπολογιών και περνάμε στο τελευταίο σημείο. Λουίς Παλοάλβες για την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κατάρτιση αυτή της γνωμοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργία των νέων Παρά το ελάχιστο διάστημα που είχα στη διάθεσή μου ήταν κάτι το πολύ προκλητικό, διότι έχουμε να κάνουμε με μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους νέους. Αυτό θα είχε δραματικές διαστάσεις για την κοινωνία στη σταδιοδρομία τους αντιμετωπίζουν την ανεργία, έχουν χαμηλότερους μισθούς και χάνουν την αυτοεκτίμησή τους κατά την κατάρτιση που λαμβάνουν. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη να μην ε, κατασπαταλήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τους νέους ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίσουν ε, τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Χάνουν λοιπόν know-how, χάνουν ε, τεχνογνωσία και σύμφωνα με το Eurofund το 2011 έχουμε να κάνουμε με απώλειες της τάξης των 153 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2013 το 23,5% των ε, νέων είναι άνεργοι με ποσοστά που κυμαίνονται από 15% στην Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, 40% στην Πορτογαλία και πάνω από 55% στην Ελλάδα και την Ισπανία. Οι ασυμμετρίες αυτές οδηγούν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας των νέων. Ήδη το 2011, 14 εκατομμύρια νέων μεταξύ 15 και 29 ούτε εργάζονται, ούτε ε, σπουδάζουν και ούτε ακολουθούν μία κατάρτιση. Πρόκειται για τους λεγόμενους NETs. Επίσης, όσοι εργάζονται, εργάζονται κάτω από επισφαλείς συνθήκες. Πώς μπορούμε να έχουμε μία Ευρώπη, πώς βλέπουμε το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τους νέους, με τον αποκλεισμό τους. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία μεγάλη μάχη κατεπηγόντως. Θα πρέπει να δημιουργηθεί βιώσιμη εργασία για τους νέους. Διαφορετικά δεν υπάρχει οικονομική δυναμική. θα πρέπει να αναλύσουμε τις ρίζες της ε, ε, κακοδαιμονίας, οι οποίες ε, σχετίζονται με διαρθρωτικά ζητήματα και εκπαιδευτικές πολιτικές που θα πρέπει να διορθωθούν. Διαφορετικά μπορεί να χαθεί μία ολόκληρη γενεά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό χρειάζονται ποιοτικές πολιτικές που να προωθούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων της οικονομίας και της κοινωνίας. Προβλέπεται ότι κάθε χρόνο 15% των θέσεων εργασίας θα ε, καταργούνται, αλλά θα δημιουργούνται αντίστοιχες. Διαφορετικά, οποιαδήποτε πολιτική απασχόλησης ε, δεν θα είναι αποδοτική. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε τρία βασικά σημεία. Μία πολιτική προοπτικών έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και κατάρτισης να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να έχουμε και μία περιφερειακή προσέγγιση όπου οι αποφάσεις να είναι πιο αποδοτικές και να λαμβάνουμε υπόψη και τα προσόντα των νέων. Να σκεφτόμαστε παγκόσμια αλλά να δρούμε τοπικά όπου η περιφερειακή διάσταση θα μας διέπει μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής προοπτικών. Επίσης θα δώσουμε ταυτότητα στο κοινό αυτό των νέων και θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθήσουν εσωτερική κατάρτιση για τους νέους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους διαφορετικά θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ κατά προτεραιότητα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα αυτή η Ευρώπη φαίνεται ότι άρχισε να κινείται. Η Επιτροπή ανακοίνωσε για τον Ιούνιο ένα πακέτο κατά της ανεργίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Μιλάμε για ένα σχέδιο εγγύηση για τους νέους που εντάσσεται στη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και καταπολέμησης του επισφαλούς χαρακτήρα απασχόλησης μέσα στα πλαίσια ενός διαθεσμικού διαπεριφερειακού χαρακτήρα, ο οποίος θα αποτελέσει χάρτη πορείας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Σε περιφερειακό επίπεδο η Γαλλία και η Γερμανία θα παρουσιάσουν ένα New Deal για την Ευρώπη για την καταπολέμηση της ε, καταπολέμησης των νέων και η ΕΤΕ θα υποστηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο κατά με 60 δις. Χρειάζονται συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως χρειάζεται και η κινητοποίηση των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κυρία Πρόεδρε, Εάν δεν υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο διαρθρωτικό και ανταγωνιστικό, τίποτα δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα εμπλεκόμενα ταμεία για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των νέων υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έτσι μόνο θα ε, καταπολεμήσουμε την πραγματική ανεργία των νέων γιατί η ανεργία των νέων απειλεί και τη δημοκρατία και την αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία μάστιγα που θα μας οδηγήσει σε μία χαμένη γενιά με μεγάλους κινδύνους μόνιμης εγκατάστασης. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Wolfgang Schäuble, ο οποίος είπε, μίλησε για μια, για μια καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιτύχουμε, διαφορετικά θα χάσουμε τη μάχη για την Ένωση της Ευρώπης. Ή ο Helmut Schmidt που μίλησε για ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει καμία, ε, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Κυρία Πρόεδρε, θα, πρέπει, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του Σκιώδης και τη Γραμματεία και το συνάδελφο Καρόνα, ο οποίος μου βοήθησε στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Είμαι στη διάθεσή σας για υποδείξεις και τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δώσουμε το λόγο στους Σκιώδης, η Βερόνικα Λόπε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του διότι σε αυτές τις χρονομοδοτήσεις δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα ιδιαίτερα σε ένα τόσο καυτό θέμα και για τη χώρα μου όπως η καταπολέμηση ανεργίας που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Θα υποβάλουμε τροπολογίες επί του θέματος και θα πρέπει να αναφερθούμε στις διαφορές και ασυμμετρίες μεταξύ περιφερειών θα πρέπει να προβλέψουμε αλλαγές και να αναθέσουμε αρμοδιότητες και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν αντέδρασαν έγκαιρα. Και πολλές φορές οι νέοι δεν είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας παρά το γεγονός ότι έχουν κατάρτιση και έχουν ε, ευρύτατη εκπαίδευση. Δηλαδή η εκπαίδευση και η παιδεία δεν ε, συμβαδίζει με την αγορά ε, εργασίας. Θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα στις χώρες όπου υπάρχει ε, ανεργία των νέων που έχει προσλάβει τόσο εκρηκτικές διαστάσεις. Η ανεργία αποτελεί μία από τις μεγάλες ανησυχίες μας και αν δεν καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Μιλάμε για ποιοτική εργασία για όλους, όμως το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι οι νέοι μας να βγουν από την ανεργία και να μπουν στην αγορά εργασίας. Ο εισηγητής θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο και με την κινητικότητα. Είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Θα πρέπει οι νέοι να μπορούν να μετακινηθούν από περιφέρεια σε περιφέρεια προς αναζήτηση εργασίας. Όμως, μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας θα πρέπει να δούμε αφενός τη θετική πλευρά, αλλά ε, οι νέοι να μπορούν να βρουν και την κατάλληλη εργασία με βάση τα προσόντα τους και να μην έχουμε διαφυγή εγκεφάλων, ε, κάτι το οποίο ζούμε έντονα στην Ισπανία. Δηλαδή οι νέοι με πολύ καλή κατάρτιση φεύγουν από την Ισπανία και μεταβαίνουν κυρίως στη Γερμανία με πολύ λίγες ελπίδες να επανέλθουν στην χώρα τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή και εδαφική συνοχή έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να εργάζονται στη χώρα τους ή στην περιφέρειά τους. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη δυναμική αυτή των περιφερειών, ιδιαίτερα των ε, ε, μειονεκτουσών. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία θα συνδράμουν σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στις ΜΜΕ. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, οι ΜΜΕ δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά για να προσλάβουν νέους θα πρέπει να τύχουν χρηματοδότηση. θα πρέπει να τις βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία αυτής της έκθεσης και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ως προς συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριε Μαδέρ δεν είναι εδώ μαζί μα. Μιράντα. Θα μιλήσω στη γλώσσα του κυρίου Άλβε και ε, Τεϊσέιρα με τα γλωσσικά λάθη που θα κάνω βεβαίως. Μιλάμε για ανεργία, για επισφαλή εργασία για ανεπίσημη και μεταβατική εργασία και εσείς μιλήσετε για ε, έλλειψη μέτρων από τις ε, κυβερνήσεις. Έτσι χάνονται ευκαιρίες για τους νέους. Στην Ισπανία και σε άλλα κράτη έγιναν μεταρρυθμίσεις, ε, δόθηκαν υποτροφίες αλλά δημιουργήθηκε αυτό το κύμα μετανάστευσης, όπως είπε και το ΕΛΚ. Έχουμε ε, να κάνουμε με μία φυγή εγκεφάλων και μιλάμε για 200.000 πρόσωπα, τα οποία μεταβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται ε, με, καλύτερη, με καλύτερους μισθούς εργάζονται στη Γαλλικία, στην Πορτογαλία και σε άλλες περιφέρειες της Ισπανίας βοηθώντας τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις και βεβαίως δεν θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι οι νέοι των μεταναστών, οι νέοι μετανάστες που δεν είναι οι ίδιοι με τους μετανάστες της Γαλλικίας ή της Πορτογαλίας της δεκαετίας του 60 και 70. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια φυγή εγκεφάλων, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκ νέου. Μιλήσατε για ασυμμετρίες. Δεν πρέπει να συγχαίουμε την κινητικότητα με τη μετανάστευση. Όταν μιλάμε για κινητικότητα, είναι άκρος ενδιαφέρουσα μέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. Αλλά δεν πρέπει να ε, διευκολύνουμε την μετανάστευση των ε, ε, εγκεφάλων του ταλέντου και να μην οδηγήσουμε σε νέες μεταναστευτικές ε, ροές των νέων. Πρόκειται για μια χαμένη γενιά την οποία θα πρέπει να ανακτήσουμε. Εμείς θα υποβάλουμε επικοδομητικές τροπολογίες για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστούμε. Σαν τη γλώσσα θα μιλήσεις, κελτικά ή αγγλικά. Χωρίς μικρόφωνο. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα πάντοτε που απαιτεί πολλά από όλους εμάς. Η ομάδα στόχος είναι οι άνεργοι νέοι που σκέφτονται ότι οι γονείς τους που τους έλεγαν να σπουδάσουν και να εξοπλιστούν ε, δεν τους βοήθησαν. Ψυχολογικά έχουν πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ιδιαίτερα στα πλαίσια του MFF, είναι αξιέπαινο αυτό. Κάποια θέματα επιμέρους τώρα. Υπάρχουν νέοι που βρίσκουν απασχόληση. Τους εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι υπάρχει υπεροπρόσφορα ε, απασχόληση εργασίας. Αυτοί ε, που τους προσλαμβάνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τους διώχνουν πριν γίνουν μόνιμοι κλπ. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζονται οι έτσι. Πολλοί πάνε σε επανειλημμένες συνεντεύξεις, σε ίντερβιου πριν πιάσουν τη δουλειά και τους αντιμετωπίζουν άσχημα. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μακριά, μακρινά ταξίδια, να δαπανίσουν ώρες για να προετοιμαστούν για το interview, να πάνε, να τους ξαναφωνάξουν για τρεις-τέσσερις ώρες, να γράψουν και κάποιες εξετάσεις και καμιά φορά μπορεί να μην τους απαντούν καν ή να τους απαντούν αγενώς. Η εταιρεία πρέπει τουλάχιστον να απαντά στους ανθρώπους ακόμα και αν δεν τους προσλάβει, να τους ε, ε, ορμηνέψει πώς θα βελτιωθούν. Αυτό θα ήταν μια ενθάρρυνση για αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους, για να μην απογοητεύονται όταν ε, περνούν από πολλές απογοητεύσεις. Γιατί όταν ε, αντιμετωπίζουν ήττα μετά την ύπα στο τέλος θα απογοητευτούν τελείως και θα απαρατηθούν ή θα πάνε να γίνουν ε, εξτρεμιστές γιατί θα στραφούν ενάντια στην κοινωνία που δεν τους φέρθηκε καλά και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Χάρηκα που μίλησε για την εκπαίδευση ο εισηγητής. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας που περιμένουν να καλυφθούν γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες στην Ευρώπη. Ε, και οι αρχές εν μέρη ευθύνονται γιατί δεν ευθυγραμμίστηκαν με την εξέλιξη της κοινωνίας, της ανάγκες των επιχειρήσεων και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να αναλάβουν πιο πολλές ευθύνες για τους αποφύτους, τι κάνουν μετά την αποφύτησή τους. Δεν μπορεί να τους δίνουν το δίπλωμα και να τους αμολάνε, για να το πούμε έτσι στον κόσμο, ε, χωρίς να ενδιαφέρονται τι θα κάνουν από εκεί και πέρα. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα περισσότερο και να τα φέρουμε σε επαφή περισσότερη με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά πρέπει να αλλάζουν επίσης συνεχώς για να λαμβάνουν υπόψη τις καινούργιες ε, ανάγκες και να είναι κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα. Από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι οι περισσότερες μιμιέ θα έλεγα παραλύουν από τους πολλούς κανονισμούς, τη γραφειοκρατία. Ε, το 20, 2020 έχουμε στόχο να μειώσουμε τη γραφειοκρατία κατά 20% και άμα γίνει αυτό θα κάνει διαφορά. Θα ενθαρρύνει τον κόσμο, θα του επιτρέψει να πάει μπροστά και να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται και αυτό είναι καλό. Τέλος, να πω ότι δεν μπορούμε μια ανοιχτή να λύσουμε το πρόβλημα. Κάποια πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη είναι θετικά και θα βοηθήσουν την κατάσταση όχι μόνο για τους νέους αλλά για όλους γενικότερα. Όπως ο κανονισμός για τις τράπεζες και τις πιστώσεις επιχειρήσεις που θα διασφαλίζονται, η ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτά θα βοηθήσουν τους νέους μακροπρόθεσμα. Τώρα, βράχει πρόθεσμα πρέπει να βοηθήσουμε να είναι αποτελεσματικές εγγύσεις για την νεολαία, να δώσει θετικά κίνητρα και αν, να, όταν ε, βρουν απασχόληση να τους ενθαρρύνουν και όχι να τους εκμεταλλεύονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Δεν ξέρω. Λουίς, θες να προσθέσεις τέλος κάτι. Ευχαριστώ. Απλώς να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που παρενέβησαν, που μιλήσαν για την κινητικότητα και τη διαφορά μεταξύ κινητικότητας και μετανάστευσης. Δεν θέλουμε να προετοιμάσουμε νέους για να μεταναστεύσουν. Θέλουμε να προετοιμάσουμε τους νέους για να ε, δώσουμε ένα νέο δυναμισμό στις ε, ντόπιε οικονομίες, σε χώριες οικονομίες και να βρούμε θέσεις εργασίας ε, διευρύνοντας και την έννοια της περιφέρειας, δηλαδή να εξεύρουμε μια εξισορρόπηση μεταξύ του νότου της Ευρώπης, διότι εδώ οι χώρες χάνουν σε οικονομική δραστηριότητα με ολέθριες συνέπειες, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε άμεσα βιώσιμες λύσεις, αλλά υπάρχουν και διαρθρωτικά ζητήματα ουσίας τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν τώρα γιατί η οικονομία εξελίσσεται και πρέπει να συμβαδίζουμε κι εμείς. Ο συνάδελφος Κέλλη μίλησε για τις καταχρήσεις που γίνονται με στοχοθέτηση τους νέους γιατί δεν υπάρχει προσφορά εργασίας παρά με ε, αμεληταίους ε, μίζερους μισθούς και τους ανατίθενται ε, καθήκοντα τα οποία, είναι πολύ, τα οποία διαφέρουν πολύ από τα πραγματικά τους προσόντα. Αυτό θα αποτελέσει ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σε βάθος Χαίρομαι και προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις, διότι νομίζω ότι κάθε υπόδειξη είναι σημαντική για ένα τόσο ε, ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μένουν ακόμα κάποιες αποφάσεις. Ε, ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. 3 Ιουνίου προτείνω, Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα. Γιατί πρέπει να σεφιστεί τον Ιούνιο. Ας κλείσουμε και αυτό το σημείο. Μένουν τα διάφορα, δεν υπάρχει κάτι από ό,τι ξέρω. Σας ενημερώνω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 19 και 20 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.